Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Άρχεται η πρωινή συνεδρίαση. Θα περάσουμε κατευθείαν Σημείο 4. Τα φυτοπροστατευτικά μέτρα κατά επιβλαβών οργανισμών. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Μάκιντάιρ. Θα ψηφίσουμε το κείμενο που έχουν συμφωνήσει τα θεσμικά όργανα που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Μάκιντάιρ. για να μας ε, μιλήσει για τη συμφωνία της 16ης ε, Δεκεμβρίου. Ο τονιστής μας, ο κύριος Άλμπερντ Ντές, έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να παρακαλέσω να έρθει να μεταφερθεί τρίτη στη σειρά των ψηφοφοριών η πρόταση κυρίας Μάκιντάιρ. Γιατί έχει καθυστερήσει και θα παρακαλούσα να της δώσουμε ένα περιθώριο να έρθει. Τι είπατε για την πρώτη ψηφοφορία που είναι τόσο σύντομη, θέλετε να τη μεταφέρουμε ή την ε, πιο εκτενή ψηφοφορία που έχουμε θέλετε να την ε, ψηφίσουμε λίγο αργότερα. Πρόεδρε, η ψηφοφορία για τις τεχνολογικές λύσεις. Καλώς. Κανένα πρόβλημα. Γίνεται δεκτή η πρόταση του κύριου Αλμπερτές. Υπάρχουν παρατηρήσεις, δηλαδή το θέμα των τεχνολογικών λύσεων θα το ψηφίσουμε τελευταίο. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Ας ψηφίσουμε λοιπόν το σημείο 6 τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπαιων. Η συγκεκριμένη μα είναι η κυρία Μίλλερ. Οπότε καλύτερα να της δώσω το λόγο. Αν το επιθυμεί φυσικά. Κυρία Μίλλερ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Βάση της ανακοινωσής μας ήταν η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον χώρο των Άλπαιων Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό εντατικά. Καλωσορίζω τη στρατηγική αυτή γιατί υπογραμμίζει την σημασία του χώρου αυτού ζωής και αναψυχής. Ευχαριστώ θερμά τους κοιόδης εισηγητές εν αναμονή των συμβαστικών τροπολογιών και γενικότερα σε όλη μας συνεργασία έδειξαν πολύ καλή διάθεση. Καταθέσαμε 11 συμβαστικές τροπολογίες και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την πρότασή μας δηλαδή υπογραμμίζουμε και τις ευκαιρίες αλλά και ιδιαίτερα τις δυσκολίε ε, του χώρου των Άλπαιων και της γεωργίας εκεί, της κτηνοτροφίας εκεί. Η δάσοκομεία, βιοτεχνία, τουρισμός και βέβαια οι γεωργικές δραστηριότητες πρέπει να προχωρήσουν ε, παράλληλα συνδεδεμένα και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε έτσι ώστε να εξασφαλίζει ο χώρος των Άλπαιων και βέβαια την, ε, φυτική, ε, την παραγωγή τροφίμων αλλά και ένα καλό περιβάλλον διαβίωσης για τους ανθρώπους. 80 εκατομμύρια σε 48 διαφορετικές περιφέρειες που καλύπτουν 7 κρατη Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, οπότε περνάμε στην ψηφοφορία. Τις συμβαστικές τροπολογίες θα τις ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε πρώτα τη συμβαστική τροπολογία 1. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ο κύριος Άγνιου. Πρόεδρε, αυτό είναι όντως διαδικαστικό. Κάποιος πρότεινε προηγουμένως να αλλάξουμε τη σειρά στον κατάλογο ψηφοφοριών. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι ψηφίζουμε για τις τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι. Ε, τι ψηφίζουμε λοιπόν. Alpines. Okay. Thank ε, κύριε Βουλευτά, ε, έπρεπε να είχατε καταλάβει από την εισηγήτρια που έκανε την παρουσίαση. Δεν καταλάβατε για ποιο θέμα μιλούσε. Συμβαστική τροπολογία 1 την ψηφίσαμε, περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην βαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε διανατάσεις της χειρός στην τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 14. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 22. Ψηφίζουμε διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 24 τώρα τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 25, 26, 27 και 28 είναι παρόμοιες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται, αλλά στο ελέγξουμε για καλό και κακό. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, Α, συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την τροπολογία 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Διανατάσσω της χειρό. Ποιο είναι υπέρ της 33. Εγκρίνεται. 37. Ποιο είναι υπέρ της τροπολογίας 37. Κατά. Απορρίπτεται. 35. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 40. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Υπάρχει πρόταση της τροπολογίας 39 και 47 και 86 να τις ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, ο και 84. Ψηφίζουμε πρώτα την 39 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ για την 39. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Την τροπολογία 47. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται και πάμε στην 84 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά Εξού και ζήτησα να γίνει ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 8. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη 42. Διανατάσσω της χειρός. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 42. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ της 53. Εγκρίνεται. 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 54. Ποιος είναι υπέρ της 54. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 55, α, συγγνώμη, τροπολογία 55, Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 58, διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ της 58. Εγκρίνεται. 63. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 64. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 69. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 74, διανατάσσω της χειρός. Ποιος είναι υπέρ της 74, εγκρίνεται. Seventy-nine. okay. 79. Πάμε στην 89 ε, λέει ο πρόεδρος, 79 μάλλον, εγκρίνεται. 80 τώρα, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 81 υπέρ, εγκρίνεται. 83, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, όπως έχει τροποποιηθεί. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Μίλλερ. Μήπως θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία εισηγητρία. Όχι, σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά. Μπορούμε τώρα... Okay. Przechodzimy do poprawki e, w takim razie do... Καλώς, σας περάσουμε στην ψηφοφορία του σημείου 7 δηλαδή την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Μπόγκοβιτς, ε, με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα δώσω και εδώ το λόγο στον εισηγητή μας, για να μας πει δύο λόγια, θα το κάνει σίγουρα καλύτερα από τον υποφαινόμενο. Κύριε Μπόγκοβιτς, έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω θερμά τους και ηγητές που κατέθεσαν μαζί με άλλους συναδέλφους 91 τροπολογίες. Είχαμε αγαστή συνεργασία, βελτιώσαμε το σχέδιο γνωμοδότησης και καταλήξαμε σε 9 συμβαστικές τροπολογίες που θεωρώ ότι καλύπτουν πλήρως όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες. Η γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότηση είναι πολύ ισορροπημένο και νομίζω αξίζει υποστήριξης. Η αρμόδια κατά ουσία επιτροπή είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας, η ΙΤΡΕ. Η δική μας γνωμοδότηση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πέθρου και στη γεωργία. Δηλαδή μιλούμε για τη βιομάζα, βιοαέριο δεύτερης γενιάς. Βλέπουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη σκοπιά της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου. Πώς θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τους στόχους μεταφοράς μας. Και επίσης ε, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. ώστε να γίνει μέγιστη χρήση του βιοαερίου στη Γεωργία και επίσης ε, ζητούμε αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και καλή σύνδεση με τα δίκτυα ώστε και το βιοαέριο να ε, γίνει εφάμιλο των υπόλοιπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πολύ σημαντική είναι η παραγωγή των ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας, γιατί δημιουργεί θέσεις απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Και καλό θα ήταν να ιδρυθούν και οι συνεταιρισμοί για να προωθηθεί η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ήπεθρο. Μιλούμε, επαναλαμβάνω, κυρίως για τα βιοκαύσιμα και την παραγωγή τους, ιδιαίτερα όταν έχουμε πλεόνασμα, χάρη στις νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και το γεωργικό εισόδημα. Ελπίζω να υπερψηφίσετε την γνωμοδότησή μου, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς την αρμόδια κατουσία Επιτροπή, την Ήτρε, για την άποψη της Επιτροπής Γεωργίας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ασθενιζόμαστε τις θέσεις σας, κύριε Σιγητά. Και φυσικά θεωρούμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, μπορούν ε, να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την αυτάρκεια της υπαίθρου σε ενεργειακά ζητήματα. Περνάμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Συμβαστική πρώτη, άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1. Τέλος ψηφοφορίας για τη συμβαστική τροπολογία 1. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογία 19. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Τέλος ψηφοφορίας. Πάμε στην 34. Ε, Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 34. Διανατάσσεως της χειρός παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 35 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44 του κυρίου Άγγινιου. Ποιος είναι υπέρ. Διανατάσσω της χειρός κατά απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στη 47 τώρα. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας ή μάλλον λάθος. 50. Τροπολογία 50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 3. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 55. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 59. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 60. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της 66. Εγκρίνεται. 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ο κύριος Μπογκόβιτς, ο εισηγητής μας παρακαλώ ζήτησε το λόγο. Στο κατάλογο ψηφοφορίας παρισέφρισε ένα λάθος για τη συγκεκριμένη τροπολογία, την υπαριθμό 5. Θα πρέπει να ψηφιστεί. Εγώ έκανα λάθος, sorry. Ε, δεν διάβασα καλά το κατάλογο ψηφοφορίας. Ήταν σωστός. Επειδή απορρίφθηκε, δεν χρειάζεται καν να ψηφίσουμε για την 5. Εγώ έκανα λάθο, λέει ο συγγητή, συγγνώμη. Ο κατάλογο ε, ψηφοφορία είναι σωστό. Τελικά τι θα γίνει με την πέντε ψηφίζουμε ή όχι. Κύριε Σιγητά, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την 5. Ογδόντα πέντε. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 86, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 87, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 4 τώρα. Διανατάσεις της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική εννέα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την εννέα. Εγκρίνεται η συμβαστική Ενέα. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης, όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Θέλετε κύριε Σιγητά να προσθέσετε κάτι. Απλώς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ε, μέριστη υποστήριξή σας και την αγαστή συνεργασία που είχαμε τους και ηγητές. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η γνωμοδότηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπράβο σας. Θα ψηφίσουμε τώρα το σημείο 4α, τα φυτοπροστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών οργανισμών. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Ανθέα Μάκιντάιρ είναι το κείμενο που αποτέλεσε το, την έκβαση των διοργανικών διαπραγματεύσεων της 16 Δεκεμβρίου του 2015, μετά από 7 τριμερείς διαλόγους που έλαβαν χώρα για το θέμα αυτό. Θα ψηφίσουμε το ενοποιημένο κείμενο που σας έχουμε μοιράσει. Η ψηφοφορία είναι ένα απλό ναι ή όχι. Αν υπερψηφίσουμε το κείμενο, θα στείλουμε επιστολή στην Ολλανδική Προεδρία με το κείμενο επισυνημένο, με την ε, στερότυπη φράση θα συστήσουμε στην Ολομέλεια την έγκριση χωρίς τροπολογίες ε, της θέσης του Συμβουλίου. Και μετά την έγκριση του κειμένου αυτού και από την Κορεπέρ και το Συμβούλιο ε, θα λάβει τη μορφή της απόφασης σε πρώτη ανάγνωση. Τη θέση σε πρώτη ανάγνωση, οπότε κατόπιν θα πρέπει να προβλέψουμε μια προθεσμία για κατάθεση των υπολογιών, προκειμένου να περάσει για την τελική οριστική έγκριση το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια. Και τώρα θα δώσω το λόγο μετά τις ε, διαδικαστικές διευκρινήσεις που έκανα εγώ στην εισηγητριά μας, την κυρία Μακεντάγερ Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ψηφοφορία, πιστεύω. Για μας, στην Επιτροπή μας, αλλά και για όλο το Κοινοβούλιο. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες. τη μέλημά μα είναι να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από διάφορα ε, ζυζάνια και φυτοκτόνα. Να δούμε μόνο την περίπτωση της ελιάς που έχει καταστραφεί από, το, από την ξυλέλα. και πρέπει να φροντίσουμε να βοηθήσουμε και να προστατέψουμε τα φυτά μας. Εδώ έχουμε προχωρήσει μέσα από πολλές διαπραγματεύσεις και αισθάνομαι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τους σκιώδεις ηγητές όλων των ομάδων που εργάστηκαν σκληρά για να ετοιμάσουμε ένα κείμενο, το είχαμε έτοιμο πριν τα Χριστούγεννα, ένα κείμενο συμβιβασμού με το Συμβούλιο υποστήριξη εκφράστηκε από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου και παρακαλώ την Επιτροπή να υπερψηφίσει αυτή τη συμφωνία σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να την εγκρίνουμε για να πάει στην Ολομέλεια το ταχύτερο δυνατό και να τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να προστατευτούν όλες μας οι χώρες από, όλα αυτά, από όλες αυτές τις αρρώστιες που απειλούν τις καλλιεργίες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας την κυρία Μάκιντάιρ. Και στο επόμενο σημείο μας ε, η συγγετρία είναι η κυρία Μακεντάιρ. Αφορά τις τεχνολογικές λύσεις για μια ισορροπημένη γεωργία, βιώσιμη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μακεντάιρ, παρακαλώ, έχετε να προσθέσετε κάτι ή θέλετε να μας εξηγήσετε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να, τυχαίνει μερικέ μερικές φορές τα πράγματα όλα να τίνουν προς την διακατεύθυνση κατεύθυνση όπως συμβαίνει εδώ. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ τους σκιώδεις όλους για την έκθεση αυτή με πολύ επικοδομητικό τρόπο συνεργάστηκαν. Ξέρουμε ότι το μέσο τη γεωργίας στηρίζεται πάντα σε νέα επιχειρησιακά μοντέλα, νέες μεθόδους παραγωγής, τεχνικές, για να βελτιώσει και την ποιότητα και την ποσότητα και να προσαρμοστεί βέβαια στις νέες και ε, καινούργιες συνθήκες. Μπορούμε λοιπόν έτσι να συμβάλλουμε στην ε, βιώσιμη γεωργία και τη διατήρηση της πρόοδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι θα μπορέσει να καταστεί πρωταγωνίστρια στην καινοτομία, την αηφορία, την ε, βελτίωση της παραγωγής. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε ένα, ζωτικό, ένα ζωντανό γεωργικό τομέα με όλες τις καινοτομίες, με τις νέες τεχνολογίες και έτσι. Για όλους βέβαια τους παραγωγούς, είτε μιλούμε για τη συμβατική, για τη βιολογική, άλλες μορφές, οι ε, κλάδους της ε, γεωργίας, θα πρέπει η καινοτομία να είναι διαθέσιμη πάντα σε όλους τους γεωργούς μας και λύσεις οι οποίες μπορεί ακόμα και σε μια μικρή κλίμακα να δίνουν καλά αποτελέσματα, ε, είναι εξίσου σημαντικές και πρέπει να προαχθούν εξίσου με αυτές οι οποίες μπορεί να δίνουν καταπληκτικά αποτελέσματα σε μεγάλη κλίμακα. Επίσης, ε, η βιοπικιλότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και υπογραμμίζεται από την έκθεση. Η γενετική ποικιλία δηλαδή πρέπει να διαφυλεχθεί και για το μέλλον. Δεν θα επεκταθώ, αλλά σας ε, παρακαλώ να υποστηρίξετε την έκθεση. Έχουμε κάνει τις ε, μέγιστες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσουμε συμβαστικές λύσεις που έχουν δεχθεί οι περισσότερες από τις ομάδες μας και ελπίζω να υπερψηφιστεί η έκθεση. Σας ευχαριστώ. Όντως, πολύ σημαντική έκθεση, δύσκολη, επίπονες εργασίες ήταν αναγκαίες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Δεκάστρο. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Μια διόρθωση, αν γίνεται. Στο άρθρο 195, τροπολογία μάλλον 195, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αντιστοιχεία με τη συμβαστική S σίγμα. Θα θέλαμε λοιπόν να ψηφιστεί ξεχωριστά 1, 9, 5. Συμβαστική S σίγμα. Ευχαριστώ. 194 και 194 ή μόνο την 195 θέλετε να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Μόνο. Μόνο την 195. Uh, yes, one, five, one, 195. Αυτή που δεν καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία Ah, e, Καλώ σα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Δεν βλέπω να θέλει άλλο κάνει το λόγο. Ή κάποιο από του πράσινου ζήτησε το λόγο. Όχι. Πάμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία Α. Άρχεται η ψηφοφορία. Ζαμέκαμ głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. 80. Τροπολογία 82 και 87. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία Β. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία Β. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83 της κυρία Κάτω. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 86. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ή e. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G. G. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορια Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 1. Συμβαστική τροπολογία... Συγγνώμη, η προηγούμενη ήταν I. Ε, συμβαστική τροπολογία J. Τέλος ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία J. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία K, K, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο, παρόλο που το είχατε προαναγγείλει. Οι 153-154 καταπίπτουν. Πάμε στην 155. Ποιος είναι υπέρ της 155? Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία M. Άρχεται ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Przyjęty. Εγκρίνεται. 166 τροπολογία τη Κάτω. ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία μη Εν. Άρχεται ψηφοφορία. Ζαμίκαμ głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία όμικρον. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 178. Διανατάσεις της χειρός. Άρχεται η ψηφοφορία. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία π. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 186, διανατάσεις της χειρός, άρχεται η ψηφοφορία. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Q. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία R. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία S. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 195. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ διανατάσεις της χειρός. Εγκρίνεται 195 και πάμε στη συμβαστική τροπολογία ΤΑΦ. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 201. Διανατάσσεως της χειρός. Παρακαλώ 201 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Σεβαστική τροπολογία U. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Sorry. Β. Συμβαστική τροπολογία Β. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 220, 21, ε, συγγνώμη. Ποιο είναι υπέρ τη 221, διανατάσεις χειρός, κατά, απορρίπτεται 221. Συμβαστική τροπολογία W, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την συμβαστική τροπολογία W. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται η W. Και περνάμε στην συμβαστική τροπολογία Χ, X. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Y. Αλλά, συγγνώμη, πρώτα την τροπολογία 228. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται 228 και πάμε συμβαστική τροπολογία Y. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Z. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΑ. Ποιος είναι. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε δύο ανατάσεις της χειρός την τροπολογία 243. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΒ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΓ. AC. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ID. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Ψηφίζουμε την 268 της κυρίας Σένερα. Ποιος είναι υπέρ, διανατάσσεται ισχυρός, χειρός, κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΕ, έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AF, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AG. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία A, A, H. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική α, 292 πρώτα, 292 του κ. Μπράνεν, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία AI, άρχεται ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 299 και 300 μαζί. Διανατάσσος της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 301. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 302 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 303. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις και αναφορές. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 και 4 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά απορρίπτεται. 6 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 9 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία AJ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 14 τώρα, της κυρίας Σκοτ κάτω. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία AK, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AL, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 της συγγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AM. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 39 της κυρίας Σένερα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία AN. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 51, 52, 53... Α, συγγνώμη. 42 πρώτα. Ποιος είναι υπέρ της 42, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία AO. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες τώρα. 51, 52, 53 μαζί. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τροπολογία 54 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55. Κατά. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κα... Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά. 59 ε, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία AP. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam Εγκρίνεται. Τροπολογία 64 της Δυνατά Διανατάσεις της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία AQ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AR. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται τροπολογία 76 της κυρίας Σκοτ Κάτω, ποιος είναι υπέρ, συγγνώμη, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 78, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και 81 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται ψηφίζουμε το κείμενο ολόκληρο μετά τις τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ για το σύνολο του κειμένου. Τέλος ψηφοφορίας. Είπα τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μάκιντάιρ. Μήπως θέλετε το λόγο. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ. Καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τους πάντες για τη συνεργασία. E, Προσοχή παρακαλώ. Ήταν η τελευταία μας ψηφοφορία. Και μάλιστα τελευταία ψηφοφορία α, για τον κύριο Βοτσεχόφσκι, τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, που ήταν στην Επιτροπή μας 12 χρόνια. Τώρα αφήνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναλάβει στο ελεκτικό συνέδριο πολύ σημαντικό αξίωμα και υπεύθυνο. Τον συγχαίρουμε θερμά. Ε, και πιστεύω ότι χάρη στην εμπειρία που έχει για τα γεωργικά θέματα θα εμπλουτίσει και την εμπειρία του ελεκτικού συνεδρίου. Ήταν ε, εισαγγελέα, δικαστής, ε, υφυπουργός, ε, πρόεδρος του είπα του Ελεκτικού Συμβουλίου στην Πολωνία και νομίζω ότι έχει όλα τα προσόντα και τα εφόδια για να αναλάβει αυτό το πολύ υπεύθυνο και σημαντικό αξίωμα στο ελεκτικό συνέδριο. Σας συγχαίρομαι κύριε Βοητσεχόφσκι, θερμά συγχαρητήρια. Μπορεί να σας ζηλεύουμε και λίγο, αλλά με μέτρο. Συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας τύχη. Panie pośle. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Σας ευχαριστώ για τα πολύ θερμά σας λόγια και σας ευχαριστώ όλους θερμά γιατί πραγματικά μου δώσατε την ευκαιρία να συναναστραφώ καταπληκτικούς ε, συναδέλφους, πολιτικούς, ε, ευρωβουλευτές ε, και με μερικούς Είχαμε δωδεκαετή πείρα ε, στην ενασχόληση με τα γεωργικά ζητήματα. Ήμουνα και αντιπρόεδρος ε, στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή αυτή και ήταν πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία που αποκόμισα για την κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την ε, ιδιαίτερη αυτή εμπειρία που είχα την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας με, κάποιο, με κάποια μικρή στεναχώρια φεύγω. Στην ακρόαση στην Επιτροπή Προπολογισμών, κατά τη γνώμη μερικών ευρωβουλευτών, ε, η εμπειρία μου ε, στην Επιτροπή Γεωργίας ήταν εμπόδιο στο έργο μου στο ελεκτικό συνέδριο, γιατί κατά τη γνώμη μερικών ε, κάποιος που ασχολείται με γεωργικά θέματα γίνεται λομπίστας ε, και δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός στον ε, έλεγχο των γεωρικών δαπανών. Αυτή ήταν η εντύπωση που δόθηκε ή αυτή ήταν η αίσθηση που είχαν μερικοί ευρωβουλευτές. Εγώ διαφωνώ κάθετα με μια τέτοια φυσικά αντίληψη και πιστεύω ότι όσοι εργάζονται και που ενδιαφέρονται ειλικρινά για την σωστή ανάπτυξη της γεωργίας ε, θα φροντίσουν για σωστή αξιοποίηση του αρκετά σημαντικού κονδύλιου της γεωργικής πολιτικής. Και μάλιστα είπα ότι εγώ στο ελεκτικό συνέδριο θα ήθελα κυρίως να ασχοληθώ με τα γεωργικά θέματα και ελπίζω να το καταφέρω, να αναλάβω αυτή την αρμοδιότητα. Και από εκεί θα σας υπηρετώ με την εμπειρία μου ε, και θα χρησιμοποιήσω αυτή την πείρα μου που αποκόμισα και από την Επιτροπή αυτή για να ε, επιτελέσω καλύτερα την αποστολή μου για το σωστό έλεγχο του, των δημόσιων κονδύλιων, των κοινοτικών κονδύλιων. Και ευχαριστώ θερμά και τον ε, κύριο Ντεκάστρο ε, που διτέλεσε και εκείνος πρόεδρος, πριν από αυτόν ο κύριος Ντόλ, ε, Νίλ Πάρης και ο με τον κύριο Ντές είχαμε πολύ στενή συνεργασία γιατί ήταν από την αρχή συντονιστή, με τον κύριο Νίκολσον, με τον Μάρκ Δαραμπέλα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τα 12 αυτά ωραία χρόνια δουλειάς και συνεργασίας που είχαμε. Πολύ σημαντική εμπειρία για μένα, ανεκτήμητη. Και θα ήθελα να σας καλέσω σε μια σύντομη αποχαιρετιστήρια δεξίωση που θα γίνει στις 6 και 4 εδώ μπροστά στην αίθουσα. Οπότε θα ελπίζω να, να τα ξαναπούμε και εκεί. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά θα έχουμε και εκεί την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσουμε και προσωπικά και να ανταλλάξουμε μερικές κουβέντες. Πάντως και εμείς πιστεύουμε, κύριε και ότι η πείρα σας από την παρουσία σας και το έργο σας στην Επιτροπή Γεωργίας θα σας βοηθήσουν για να επιτελέσετε και στο ελεκτικό συνέδριο καλύτερα τη λειτουργία και το αξίωμά σας. Και μάλιστα είχαμε πολύ αγαστή συνεργασία με το ελεκτικό συνέδριο. Ελπίζω να, γίνει σωστή, να συνεχιστεί ο σωστό έλεγχο των γεωρικών δαπανών. Σα ευχαριστούμε, Σα χαίρουμε και πάλι θερμά και ραντεβού στι 6 και 4 για το κοκτέιλ. Αλλά μέχρι τις 7 Μαΐου θα εξακολουθείτε να είστε μέλος της Επιτροπής. Μέχρι τότε θα σας έχουμε κοντά μας, μετά θα αναλάβετε. Ο κύριος Άγνιου. Είναι καλή ευκαιρία νομίζω να ρωτήσουμε τον κύριο Βουιστσαχόφσκι εάν ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου θα ήταν διατεθειμένος να επισκεφθεί κάποιες από εκείνες τις χώρες όπου δαπανώνται υπερβολικά πολλά υψηλά ποσά για την ανάπτυξη της υπαίθρου και να φροντίζει να χτίζονται τα κτίρια για τα οποία δίνουμε τα λεφτά και αν χτιστούν να πηγαίνει και κάποιος να δουλεύει εκεί μέσα γιατί χτίστηκε νομίζω ένα κέντρο στην Ουγγαρία ως τάχα διοικητικό κέντρο για τα κακοποιημένα, κακοποιημένα σκυλιά ε, και τελικά ούτε καν άνοιξε τις πόρτες του. Ξέρετε ότι η πατρίδα μου, το Ρωμανό Βασίλειο, προσφέρει χρήματα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ω καθαρό χορηγό και δεν είμαστε τεθειμένοι να ανεχθούμε κάτι τέτοιο περισσότερο να συμβαίνει. Είστε λοιπόν τεθειμένο να πάτε και να τα κάνετε όλα λαμπίκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά είχατε την ευκαιρία τέτοιε ερωτήσει να τις θέσετε στην ε, ακρόση που έγινε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού για τη θέση αυτή στον κύριο Βατσεχόφσκι. Τότε έγινε η ακρόση, τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή να τεθούνται τις ερωτήσεις και να ληφθούν απαντήσεις. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για τέτοια συζήτηση. Στην επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βοητσεχόφ και όταν θα έρθει με την ιδιότητά του ως μέλος του ηλεκτρικού συνεδρίου, τότε θα του δώσουμε, ίσως θα έχουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε τις ερωτήσεις. Να με συμπαθάτε κύριε Άγνιου, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή για την ερώτηση αυτή τώρα. Στο μέλλον, το θα έρθει ως μέλος του ηλεκτρικού συνεδρίου, μπορείτε να την υποβάλλετε. Παρακαλώ. Ζητήθηκε αναβολή προς το παρόν του σημείου 10, γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να έρθουν εγκαίρως, υπήρχε πρόβλημα με τις πτήσεις. Ε, για την μακρόπνοη και καινοτόμα στρατηγική στην εμπορική και επενδυτική πολιτική, ε, η κυρία Δεράς Γκαρσία που δυστυχώ απουσιάζει. Η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου είναι αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή. Αντικαθιστώντας την κυρία Δεράς Γκαρσία θα λάβει το λόγο ο κύριο Μισελ Νταντά. Χαιρόμαστε για την ενασχόληση με το θέμα αυτό, γιατί κατά τη γνώμη μου οι εμπορικές συμφωνίες που εξετάζονται αυτή τη στιγμή δεν ε, λαμβάνονται όντως ε, υπόψη τα συμφέροντα των Ευρωπαίων γεωργών και εμπόρων. Αυτά θα τα πούμε και στη συζήτηση με τον Αρμόδιο Επίτροπο. Πάντως, η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι εμπορικές αυτές συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση δεν εξετάζουν δεόντως τα αποτελέσματα που θα έχουν στη Γεωργία. Και γίνεται μια πολιτικοποίηση της συζήτησης και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε χειρό μήνυμα εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας. Αλλιώς ε, θα εκτεθούμε στις επικρίσεις και τις μορφές των γεωργών στο μέλλον, γιατί δεν προασπίσαμε δεόντως τα συμφέροντά τους. Και θα έρθουμε στο σημείο που βρισκόμαστε και απέναντι στην ε, κοινή γεωργική πολιτική. τώρα μας κατηγορούν ε, για μερικές συνέπειες της κοινής γεωργικής πολιτικής, ε, ενώ εμείς συμμετείχαμε στην εκπόνηση της όταν συμφωνήθηκε ένα προσωπικό σχόλιο λοιπόν και ζητώ συγγνώμη που παρέτεινα κάπως τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νταντάν που θα παρουσιάσει την έκθεση της κυρίας Εράνς Γκαρσία. Συγγνώμη. Θα σα διαβάσω την ε, επιστολή τη συναδέλφου, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, το συγγνώμη για την αποσία τη κυρία Έρανς που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας για λόγους ανεξάρτητους της ελευθερήσεώς της. Με παρακάλεσε να παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης για μια νέα και καινοτόμο στρατηγική μακρόπνοη για το εμπόριο και τις επενδύσει στο μέλλον. Ε, για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τις κρίσεις τη γεωργίας θα πρέπει και να κατακτηθούν νέα μερίδια αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και έξω από τα σύνορά μας. Υπό την προπόθεση βεβαίως ότι θα εξασφαλίζεται κατάλληλη η προστασία των πιο ευάλωτων τομέων και ότι θα αποφεύγεται ιδιαίτερω η μετατροπή τη γεωργία σε συναλλαγματική ισοδύναμη όπω έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Απαραίτητο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει κατά τρόπο συστηματικό και σοβαρό στην αξιολόγηση των συνεπειών για πιθανέ ε, συνέπειε σε τρίτε χώρε και αυτέ οι μελέτε να διαβεβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την έγκριση ή απόρριψη εσδήποτε εμπορική συμφωνία. Οι συμφωνίε εμπορικέ που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προτείνουν συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των ε, ε, εταίρων ε, με συνθήκες βεβαίως περιβάλλοντος, κοινωνικές συνθήκες, περιβαλλοντικές συνθήκες πάρα πολύ αυστηρές, τις αυστηρότερες του κόσμου. Τέτοια λοιπόν ισότιμη αντιμετώπιση μέσα από αυτές τις εμπορικές συμφωνίες θα διευκόλυνε τον Ευρωπαίο παραγωγό και γεωργό να αξιοποιήσει περισσότερο τα ανοίγματα νέων αγορών όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών προελεύσεων η θέση μας πρέπει να είναι άτεγκτη κατά την σύναψη συμφωνιών με τρίτα κράτη, ιδιαίτερως δε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ονόματα προελεύσεως και οι γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τα, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κοινής πολιτικής, γιατί έτσι καθιστούν ορατές τις προσπάθειες ποιότητας που έχει αναλάβει ο Ευρωπαίος παραγωγός. Και γι' αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων που απειλούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τα φυτογεινά ε, φράγματα προστασίας θα πρέπει να εξασφαλιστεί σημαντική πρόοδος ώστε τα ε, εμπόδια, ε, τα αδικαιολόγητα και οι φραγμοί που αφορούν τις εξαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων θα να καμφθούν χωρίς βεβαίως να υπάρξει ουδεμία υποχώρηση σε σχέση με τα θέματα δημόσιας υγείας και καταναλωτού. Πρέπει επίσης να δώσουμε χώρο σε σχέση με την δυνατότητα έκφρασης μέσα από γνωμοδοτήσεις, πρέπει να υποστηριχθεί βέβαια η κύρια έκθεση, οι δεσμεύσεις οι δασμολογικές ε, που επιβάλλονται στη βάση με, τρίτους, με τις τρίτες χώρες ε, πρέπει να εξεταστούν. Έχουμε 71% των γεωργικών συμβάσεων συναλλαγών σε γεωργικά προϊόντα με μηδενικούς δασμούς, ωστόσο πρέπει να έχουμε ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο με υποστήριξη ιδιαίτερως της διάστασης της ανταγωνιστικότητας υπέρ των ε, εξαγωγών, της βελτίωσης παραγωγής και του ανοίγματο προς τις ξένες αγορές. Θα πρέπει να προβλεφθεί και η βελτίωση της ε, γεωργικής παραγωγής για να ανταποκριθεί ε, αυτή στην ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού και βέβαια τις κλιματολογικές αλλαγές. Για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν εκστρατείες ενημέρωσης, φιλόδοξες, ευφύης, με υπογράμμιση τίτερα των προϊόντων, με προβολή των προϊόντων μας, τόσο μέσα όσο και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε το χειρότερο δυνατό να δούμε τα αποτελέσματα για την προογή των Ευρωπαϊκών γεωργικών γεωργικών προϊόντων που η κυρία Ράντσα Γκαρσία επεξεργάστηκε πέρσι και που θα μπορούσε να έχει τεράστια ανταπόκριση, απήχηση ω προ την προβολή. Αυτά είναι τα στοιχεία που θέλω να υπογραμμίσει συνάδελφο, αγαπητοί συνάδελφοι, με παρακάλεσε να σας διαβιβάσω την διάθεση και βούλησή της να δεχθεί στο δυνατόν περισσότερα σχόλια και βεβαίως ε, τις ευχαριστίες της προς όλους αυτούς που την υποστήριξαν στη δουλειά αυτή και βέβαια πρόεδρε θα σας δώσω και εγώ το λόγο μετά για να κάνω τα προσωπικά μου σχόλια. Μάλιστα. Συζήτηση τώρα. Χρόνο έχουμε, οπότε θα είναι πολύ αυστηρός στην τήρηση του χρόνου μιλίωση. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ναι. Κύριο Βιέγα είναι ο σκιώδη, δεν μπορεί όμω δυστυχώ να είναι εδώ. Έτσι έχω και εγώ κάτι να σα διαβάσω αν δεν έχετε αντίρρηση. Μπορώ. Ευχαριστώ. Η έκθεση περιλαμβάνει θετικέ πτυχέ και υπογραμμίζει εύστοχα κάποια αίτια που και εμεί ε, εντοπίζουμε, ωστόσο δεν καλύπτει επαρκώ όλε τι πτυχέ που πρέπει να συζητηθούν στο σημείο 3. Ο κύριος Βιέγκας ε, σημειώνει ότι πρόκειται για έκφραση μιας αφέλειας γιατί ε, όταν μιλάει για παγκόσμιο ε, εμπόριο δεν επισημαίνει τα προβλήματα της TTIP που μας απασχολούν εδώ και χρόνια. Εδώ υπάρχει ένα ανώτατο όριο που έχει επιβληθεί για τα εισοδήματα των ε, γεωργών, οι συμφωνίες της ΓΑΤ ε, από το 1947, αλλά ιδιαίτερα μετά το 1996 και το γύρο της Ουρουγουάης έχουν καταβαραθρώσει το, ε, τους γεωργούς της Ευρώπης. Έχει χαθεί το ιδιαίτερο καθεστώς του οποίου έχεραν και πρέπει να προχωρήσουμε με μια κοινωνική συνοχή, η οποία τώρα έχει λησμονηθεί, όπως και η εδαφική. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, παρακαλώ πιο αργά. Πιο αργά μας ακούτε. Και θα μπορούσε έτσι να ε, διαπραγματευτεί ε, ίσους όρους στις διεθνείς αγορές. τα όσα είχαν προβλεφθεί λοιπόν ε, για συζήτηση δεν έχουν συζητηθεί όπως θα έπρεπε. Αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να στηριχθούμε μόνο στο απελευθερωμένο εμπόριο και τις αρχές της, αγορά, της ζήτησης και της προσφοράς. Ε, η ιστορία θα αποδείξει ότι θα ήταν κάτι τέτοιο πάρα πολύ μεγάλο ε, ε, λάθος. Έχουμε την αρχή της πρόληψης, έχουμε την αρχή των γεωγραφικών ε, ονομασιών προελεύσεως Έχουμε προσπάθειες για ε, προστασία της βιοποικιλότητας, για αποτροπή της απερίμωσης και δεν μπορούμε να, ταχθούμε σε τόσο, ε, να υποταχθούμε σε τόσο μεγάλη πίεση και για το περιβάλλον και για, τα, για την κοινωνική διάσταση και τη γεωργία μας όπως αυτό που απαιτεί τη TIP. Δεν θα επιτρέψουμε να υποβαθμιστεί περαιτέρω η γεωργία μας και σας ευχαριστώ. Η διερμηνείς σας να μιλάτε με πιο φυσιολογικό ρυθμό για να μπορούν να σας παρακολουθούν και διερμηνείς και να μεταφέρουν τα μηνύματα και τις σκέψεις σας. Ο κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω με λίγα λόγια πόσο συμφωνώ με την κυρία Χεράμις Καρσία για αυτή την έκθεση συγκεκριμένα. Ιδίω όταν μας λέει ότι η γεωργία θα πρέπει να προσαρμοστεί. Αλλά όχι μέσω του, της πλειοδοσίας του παζαρέματος με τις πολυεθνικές, με τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Ο κλάδος της γεωργίας είναι στρατηγική σημασίας και ξέρουμε εδώ ότι διακυβεύονται η διαφύλαξη της επιστημικής μας ασφάλειας και του δυτικού μας επίπεδου και το λέω με πυγμή, δεν θέλουμε να συναυθεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Το λέμε διαρκώ. Η Γεωργία πρέπει να ξαναμπεί στην καρδιά των διαπραγματεύσεων. Για όσα υπόθηκαν, να θυμίσουμε ότι η συμφωνία πρέπει να είναι ισόρροπη σε όλα τις τα συστατικά στοιχεία, είτε δασμολογικά είτε μη δασμολογικά, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και για τη μέγιστη δυνατή σύνεση σύνεση στις προσθήκες που θα γίνουν στην έκθεση για, την πρόσβαση στην αγορά. Πρέπει να, να προστατεύσουμε τα πιο ευπαθή ε, κομμάτια της γεωργικής αγοράς, ιδίως στην περίοδο που διανύουμε. Ο κλάδος αυτός είναι σημαντικός για την προσφορά θέσεων απασχόλησης, ιδίως στις περιοχές με τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα. Η προστασία αυτού του ευαίσθητου κλάδου θα καθορίσει τις συνολικές μας στρατηγικές αυτές που εφαρμόζουμε σε όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες. Γι' αυτό πρέπει να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε μια συνολική θεώρηση όλων των συμφωνιών που αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης. Διότι δεν μπορούμε να παραχωρούμε ανεξέλεγκτα ανταλλάγματα. Και για τα υγειονομικά και φετογειονομικά ε, θέματα, για όλα τα θέματα της επιστικής ασφάλειας, θα πρέπει να μην υποβαθμίσουμε τις νομοθετικές μας προβλέψεις, να μην ε, διαταραχθεί η αρχή της προφύλαξης και κυρίως να προστατεύουμε τους πολίτες και τους καταναλωτές. Επίσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ένα μείζον κεφάλαιο στις συμφωνίες που συζητούμε αυτή τη στιγμή με ΗΠΑ, δεν πρέπει να υποχωρήσουμε ούτε σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να προστατεύουμε τις διαφορετικές μας ενδείξεις και να τις προστατεύουμε από την πειρατεία και τις παρατήσει και για το καλό των επιμέρου περιοχών και για του καταναλωτέ. Πρέπει να αρνοθούμε, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, θα την περιλάβω σε μια τροπολογία, οποιαδήποτε σύναψη εμπορική συμφωνία που δεν σέβεται τι γεωγραφικέ ενδείξει. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ όταν ε, ξεπερνάτε τον χρόνο μιλία να μην υπερβάλλετε κιόλας. Κυρία Νόχη, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Με ενδιαφέρει στο σημείο 3 και 4 η ε, αναφορά στους δικούς μας γεωργούς βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε τα δικά τους συμφέροντα. Όταν όμως έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα με ροές μεταναστευτικές από ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να μιλούμε όχι μόνο για την αξιολόγηση των συνεπειών για τους δικούς μας γεωργούς, ε, γιατί ε, επηρεάζονται από τα προβλήματα τα κλιματικά και τα λοιπά προβλήματα όλοι οι γεωργοί στον κόσμο. Εάν νομίζει κανείς ότι μπορούμε εις βάρος των άλλων να κερδίζουμε, να κάνουμε ε, καλές ε, δουλειές, τότε δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όλων αυτών των ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύουν από τη μια περιοχή του κόσμου στην άλλη. Ευχαριστώ Νίκολσον. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σωστό όρισε ως προτεραιότητά της το διεθνές εμπόριο και, και, του αναγνωρίζει τη σημασία του και η δική μου βέβαια κυβέρνηση αλλά και όλοι οι παραγωγείς σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν σε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίθεση μεταξύ του ελεύθερου και του δίκαιου ή ισοδίκαιου εμπορίου. Ε, βέβαια Πρέπει να κοιτάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει το στόχο του δικαίου εμπορίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ερικέ φορέ ίσω μόνο ω διαπραγματευτικό επιχείρημα μπορεί να προβάλλεται. Και όπω είπα και στην Ολομέλεια κάποια στιγμή, έχουμε από τη μια τον Επίτροπο Χόγκανο ο οποίο προσπαθεί να γύρει και να υποστηρίξει ζητήματα συμφερόντων των γεωργών που χάνουν χρήματα μέσα στην Ευρώπη από τις γεωργικές της δραστηριότητες, ενώ η Επίτροπος Μάλστρομ ε, έχει πάρει τους δρόμους και γυρνάει σε όλο τον κόσμο για να αναπτύξει νέες αγορές, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από αυτό το άνοιγμα. Η TTIP, η σχέση μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, νομίζω μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες για ευάλωτους ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τομείς, κυρίως το βοδινό και τα γαλακτοκομικά και είναι μεγαλύτερη ακόμη η κίνδυνα αν προχωρήσουμε σε περισσότερη απελευθέρωση. Εάν οι μη δασμολογικοί φραγμοί καταργηθούν, κάθε τομέα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας θα χάσει από ε, από κάθε τομέα λοιπόν θα χάσουμε, εκτός ίσως από τα οπορικά. Ανεξαρτήτως δε των συνεπειών των ε, εκλογών σε μένες πολιτείες και δεν θα σχολιάσουμε εδώ πέρα το αν ο κύριος Τραμπ μπορεί να ε, γύρει τείχος ή ποιος θα ήταν ο καλύτερος υποψήφιος ως πρόεδρος της ΗΠΑ για την Ευρώπη. Πάντως η DTIP δεν πρόκειται να μας ε, δεν πρόκειται να λύσει προβλήματα. Του αντίον θα την έχουμε κοντά μα για αρκετό διάστημα και τα σχετικά προβλήματα. Η Μερκασούρ επίση είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να κοιτάξουμε, διότι η παραγωγή βοη κρέατο ε, εκεί είναι τέτοια, τέτοιο μέγεθο σε τέτοια μορφή που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να την ανταγωνιστούμε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δηλώνει πως είχε αρχικά προτάσεις για δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τόνους βοδινού που θα σήμαιναν ότι θα κατακλυζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να που φαίνεται τώρα ότι η Ευρώπη δέχεται ήδη αυτήν την ε, εισαγωγή. Αυτή φαίνεται, ε, αυτές τις εισαγωγές, αυτή φαίνεται να είναι η εντύπωση τουλάχιστον στον πολίτη και τον κτηνοτρόφο πάνω απ' όλα. Και, πάνω, και πρέπει να φροντίσουμε να καθησυχάσουμε τους γεωργούς μας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ. Και εγώ πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν παρκή δραστηριότητα, αλλά και θα έπρεπε και οι γεωργοί μας να δραστηριοποιηθούν. Ο κύριος Φεγάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για να συμπληρώσω όσα υπόθηκαν, με τα οποία συμφωνώ απολύτως. Απλώς να πω ότι στο πλαίσιο τη κρίση και της λιτότητας, στο οποίο έχουμε βυθίσει του Ευρωπαίους Γεωργούς, Καλό θα ήταν να καταγγείλουμε σε αυτό το σώμα το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βοηθά γεωργού άλλων χωρών που δεν είναι μέλη τη Ένωση. Μιλάω για τη Μολδαβία, που πήρε τελωνιακή βοήθεια για να στηρίξει την κεντρική τη παραγωγή, θύμα του ρωσικού εμπάρκου και την Τινησία που πήρε στήριξη για τα προκυπευτικά τη. Όμως, αυτό που με ενοχλεί κυρίω είναι το γεγονό ότι η Τινησία σήμερα, που είναι ένα μεγάλο ανταγωνιστής για την Νότια Ευρώπη, δεν σέβεται καν του κανόνους μα. Ιδίω μα απρέκυψαν για το κεράσι. Και το γνωστό φυτοφάρμακο Ντιμιτοάτ. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε κυρίως τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε, κυρία Τζοφίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση που θίγει τα βασικά θέματα των σχέσεων μεταξύ γεωργίας και διεθνούς εμπορίου. Θα ήθελα να σταθώ στα σημεία που θεωρώ εγώ κρίσιμη σημασία και θέλουμε να τους δώσουμε έμφαση για να τα εξετάσει μετά και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Η γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής ήταν καθοριστική σημασία και αυτό το δείχνει η άποψη ότι, αυτό το δείχνει το γεγονός ότι στην καθήλυνη στην έκθεση της καθέλην αρμόδιας συγκήτριας. Μιλάμε πολύ συχνά για, την, ε, για τις εμπορικές διαστάσεις, αλλά όχι για τη γεωργία. Αυτό λοιπόν ε, δείχνει ότι πρέπει να δείξουμε πυγμή και να είμαστε πολύ σαφείς στα μηνύματά μας. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι η γεωργία ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ε, ένα νόμισμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγορά ισοτιμιών. Θα πρέπει οι διεθνεί αγορέ να ανοίξουν και να δοθούν μεγάλε ευκαιρίε στου γεωργού, αλλά μέσα από πολυμερεί διμερεί συμφωνίε, εφόσον οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν μηχανισμούς αμοιβαιότητας και ειχνηλασιμότητας των προϊόντων. Αυτοί θα πρέπει να επιτρέπουν στον καταναλωτή να διαπιστώσει την πραγματική τους προέλευση και κατά συνέπεια και τις μεθόδους καλλιέργειας που έχουν χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην πραγματική αντιστοιχεία των φυτογενομικών μας μέτρων και διατάξεων. Θα πρέπει να δούμε τι υποχρεώσεις βαρύνουν τους Ευρωπαίους γεωργούς ε, ως προς την ε, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την επισητιστική ασφάλεια εφόσον δεν εφαρμόζονται στην πράξη και κάποιες φορές ε, προϊόντα που έρχονται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνίζονται τα δικά μας τα προϊόντα. Αυτό το, τονίζει έτσι καλώς και η συγκήτρια. Θα πρέπει να έχουμε και δυσφαλιστικά μέτρα, τα οποία να μπορεί κανείς ε, πραγματικά να τα επικαλεστεί και με μηχανισμούς εξέτασης πιο ευέλικτους, που να μην είναι μόνο επί χάρτου διατάξεις. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της ντομάτας ε, συμφωνίες, οι οποίες παραμένουν στην αιγίδα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μόνον, αλλά τελικά δεν ενεργοποιούνται ποτέ. Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Αγορά δεν μπορεί μόνο να αξιολογείται συνολικά. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στις επιμέρους αγορές, τις τοπικές αγορές, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπος. Έτσι και οι μελέτες αντικτύπου θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές και ακριβείς, δίνοντας ε, το την απαραίτητη έμφαση στην τοπική και περιφερειακή διάσταση, είτε εξάντια κατά τη διάρκεια εφαρμογής των συμφωνιών. Αυτό είναι ένα σημασία σημείο που το είδαμε και με την έκθεση που εγκρίναμε ε, σχεδόν ε, τυφλά. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ενημέρωσης αλλά αυτή θα πρέπει να μα δίνει μια διαρκή και, καταλα... και λεπτομερή επισκόπηση για τι εμπορικέ ανταλλαγέ, Διότι εφόσον τα εμπορεύματα δεν ανοιχνεύονται δεν είναι ε, σωστό το σύστημα. Και θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα για την προστασία και τη διασφάλιση των γεωγραφικών ενδείξεων ε, σε όλες τις εμπορικές συμφωνίε των οποίων το TTIP δεν είναι μια καλή περίπτωση. Ευχαριστούμε κυρία Μακίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία για αυτή την ε, έκθεση έξι εδαφείων. Θα... Πρέπει να θυμάμαστε ότι η Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Για αυτό ό,τι θα πούμε θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί και πάρα πολύ ακριβεί. Θα πρέπει το ε, Κοινοβούλιο να θυμάται τι έγινε με τον Πέτρε Μάντελσον όταν ε, είχε την ε, γνωμοδότησε για τις συμφωνίες διεθνού εμπορίου ε, που μας αγνόησε και ε, τις προειδοποίησεις δεν τις λάβαμε προσεκτικά υπόψη. Το είδαμε από διμερεί συζητήσει στη συνέχεια. Ποιε ήταν οι επιπτώσει. Με ενδιαφέρει λοιπόν ακριβώ αυτό. Ποιο ήταν ο αντίκτυπο των διαφόρων ε, διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Είμαι υπέρ του εμπορίου. Αλλά η θέση τη Γεωργία για πολλά ε, κρατημέλη είναι πραγματικά ευαίσθητη και είναι διαφορετικέ οι καταστάσει ανάλογα με τα διάφορα προϊόντα. Η Μερκοσούρ είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για τον τομέα του βόη, όπω είπε και ο κ. Νίκολσον. Μπορεί να είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και στι συγκεκριμένε επαρχίε μα. Από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε, να έχουμε επίγνωση των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να προκαλέσει μια συμφωνία. Και πραγματικά ως Επιτροπή Γεωργίας θέλουμε να μιλήσουμε στους συναδέλφους μας των εμπορικών υποθέσεων για να καταλάβουν τις δικές μας ευαισθησίες, τα ευπαθή σημεία και να τα λάβουν υπόψη. Να μην δώσουν ως αντάλλαγμα τη γεωργία μας, να προστατεύσουμε τα ευπαθή προϊόντα με τον καλύτερο τρόπο. Διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργία αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Κατά την άποψή μου είναι σημαντική αυτή η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σωστά μιλήσατε για σόρευση αποτελεσμάτων. Γιατί ε, μια παραχώρηση από εδώ, μια παραχώρηση από εκεί, από τα μικρά αυτά ρεύματα δημιουργείται ένας ε, πολύ ορμητικός σχήμαρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σελίμωβιτς. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πολύ καλή η γνωμοδότηση στη διατύπωσή της ε, με κάποιες διαφοροποιήσεις ίσως θα μείνουμε πιστοί στο πνεύμα θεωρούμε ως φιλελεύθεροι ότι το εμπόριο είναι θεμελιώδης αξία χωρίς αυτό δεν, μπορούμε να, δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία του του πιστεύουμε ότι η γεωργία παρά εξετέθη ως διαπραγματευτικό χαρτί σε διαπραγματεύσεις εμπορικές. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό ή δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κατά τρόπον ώστε να προβάλλεται η Γεωργία στο μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί σε διαπραγματεύσεις. Γιατί βεβαίως κάθε τι μπορεί να αποτελέσει ένα επιχείρημα ε, άσο στο μανίκι, αλλά δεν πρέπει πάντα να είναι αυτό η γεωργία. Ιδιαίτερα θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία των διαπραγματεύσεων της DTIP, της ολοκλήρωσης τους και πάνω από όλα της εξασφάλισης ενός τρόπου ισοδίκαιου και ισορροπημένου για να εξυπηρετηθούν και τα συμφέροντα της γεωργίας και των γοργών. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ζημία που έχει φέρει η απουσία εμπορίου από το γεωργικό τομέα ήταν πολύ σημαντική και ιδιαίτερα βλέπουμε τις αρνητικές συνέπειες του ρωσικού εμπάργου στον γεωργικό τομέα της το άνοιγμα λοιπόν νέων αγορών αποτελεί σημαντική ευκαιρία και διέξοδο, ευκαιρία διεξόδου από τη γεωργική κρίση στο μέσο της οποίας βρισκόμαστε. Αλλά πρέπει ιδιαίτερα να σημειώσω ότι δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε στην ψευδέστηση ότι μια εμπορική συμφωνία μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα του γεωργικού τομέα. Πρέπει ο γεωργικός τομέας ο ίδιος να δώσει απαντήσεις στα προβλήματά του. Και βέβαια ένα μέρος αυτών των λύσεων θα είναι το άνοιγμα καινούριων αγορών. Ευχαριστώ θερμά. Το θέμα είναι πώς θα εξυγχρονιστούμε και προς ποια κατεύθυνση. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Στο θέμα του συναλλαγματικού χαρτιού βεβαίω και του σοβαρού επιχειρήματο δεν θα επανέλθω, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα στον τομέα την αξία του τομέα με τις ιδιαιτερότητες του ε, και βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μπορεί να καθίσατε και πιο ευάλωτος λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Γι' αυτό θα ήταν καλό να εξασφαλιστεί η να δυνατόν πιο επικαιροποιημένη, πιο ε, ισορροπημένη συμφωνία. Πρέπει να κοιτάξουμε τους κύριους εταίρους μας ε, και ανταγωνιστές, Ηνωμένες Πολιτείες όπως αναφέρθηκε, Μερκοσούρ, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία πολύ σύντομα οι ανταλλαγές λοιπόν ε, με απαλλαγή τελωνιακών δασμών με την Mercosur δεν είναι ασφαλής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με συμφωνίες του 2004. Κατά λέξη έχουν αντιγραφεί, ενώ το μεταξύ έχει αλλάξει τόσο πολύ ο κόσμος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει ιδιαίτερα να ε, επαγρυπνεί σε σχέση με, τα σορευτικά με τις σωρευτικές συνέπειες αυτών των ε, συμφωνιών και βέβαια πρέπει να προσέξουμε και τις εμπορικές πρακτικές και τις συνέπειες κοινής γεωργικής πολιτικής όπως την προβλέπουν οι συνθήκες σταθεροποίησης λέει, της αγοράς και του γεωργικού εισοδήματος. Δεν μπορούμε από τη μια να στηρίζουμε τους γεωργούς μας με τον προπολογισμό της ΚΑΠ που όλο και μειούται και ταυτόχρονα να τους εκθέτουμε στην, στον των ανταγωνισμών των πιο ανταγωνιστικών περιοχών του κόσμου στον τομέα, στον τομέα της γεωργίας. Επίσης, δεν πρέπει να λησμονούμε τις πολυμερείς συμφωνίες. Ε, Στον Αράουι έγινε πρόσφατα ο νέος γύρος συνομιλιών ε, της, ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Δεν μπορούμε να λησμονούμε τα προβλήματα του γεωργικού κόσμου στις διαπραγματεύσει αυτές και ρωτώ για άλλη μια φορά εάν έχει εκπνεύσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Εγώ θεωρώ πως δεν υπάρχει πια, απλώς παραμένουν κάποιες δικαιοδοσίες του. Έτσι λοιπόν... Με τον νέο αυτόν γύρο πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της έναντι του ΠΟΕ και να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν τον τελευταίο ναήτη υπότι στην, ε, με την παραχώρηση ε, όλο και πεστούρα εδάφους από τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν εγκαταλείψει τον ΠΟΕ. Πρέπει εμείς άραγε να συνεχίσουμε να τον υπερασπιζόμαστε και να εφαρμόζουμε τις αρχές του. Ευχαριστώ. Πολύ συχνά μάλιστα να λαμβάνουμε και πρωτοβουλίες εμείς από μόνοι μας στον ΠΟΕ. Και έτσι εκθέτουμε τη θέση μας. Ο κύριος Έρντος. Csodálkozom, hogy az Európai Bizottság hatásvizsgálatok nélkül próbálja megnyitni az Európai Unió. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ η ανάλυση, η μελέτη αντικτύπου, όπως είπε και ο συνάδελφος Νίκολσον, δείχνει ότι έχουμε 78 τόνους βόηου κρέατος και επίσης 70 τόνους πουλερικών, 100, 700 μάλλον τόνους καλαμποκιού και 750 τόνους ε, εθανόλης που έρχονται προς την Ευρώπη. Αυτά θα συμβούν. Μπορείτε να μας πείτε πόσες μικροεπιχειρήσεις της Ευρώπης, πόσοι γεωργοί θα πτωχεύσουν εξαιτία αυτών των ε, γεγονότων. Ευχαριστούμε κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που οι συνάδελφοι Μαγκίνες και Νίκολσον έθιξαν το θέμα της Μαρκοσούρ. Κατέδειξαν ορθώς ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση και διαπραγματευτεί με αυτές τις νοτιοαμερικανικές χώρες θα προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες για την βιομηχανία βόηου στην Ιρλανδία και προφανώς και στην Βρετανία. Η Μαρέιτ Μαγκίνες είναι από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και ο κύριος Νίκολσον από τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό καλύπτει όλη την ίσο της Ιρλανδίας με ένα πολύ ζωντανό ε, ζωικό κεφάλαιο που μπορεί όμως να πληγεί από τις εισαγωγές από την Αργεντινή λόγου χάρη. Παρόλα αυτά, αν το χρησιμοποιήσω αυτό σε επιχείρημα στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα, οι Γεωργοί δεν καταλαβαίνουν τι του λέω, γιατί πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει το σωστό. Δεν είναι όμω έτσι. Όλοι μας που εκπροσωπούμε περιοχές όπου υπάρχουν βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο, θα έπρεπε να καταδικάζουμε αυτά που συμβαίνουν στην Μερκοσούρ. Όμως, δεν ε, ε, διαπραγματευόμαστε τη συμφωνία TTIP με τη Μερκοσούρ. Έχω περάσει έξι ώρες σε, δύο διαφορετικές, σε πολλές διαφορετικές συναντήσεις στην αίθουσα των για να μιλήσω με τους υπεύθυνους της Γεωργίας ε, στη, της TTIP. Και αναρωτιέμαι εάν οι συνάδελφοι ε, της ε, Επιτροπής Γεωργίας έχουν πάει και αυτοί στο αναγνωστήριο που διατίθεται τα κείμενα της Συμφωνίας TTIP για να δουν αυτά που έχω δει και εγώ με τα μάτια μου. Ευχαριστώ. Κύριε Άγνιο. Οπότε, υπολογίζουμε σε εσά ε, όταν είναι εδώ ο Επίτροπος και έχουμε τη σχετική συζήτηση, υπολογίζουμε σε εσά να υψώσετε τη φωνή σας και να θέσετε τις σχετικές ερωτήσεις. Ο κύριος Γιάρ. Πρέπει να ομολογήσω ότι και εγώ πολλές φορές πήγα στον αγνωστήριο και διάβασα τα κείμενα για τη γεωργία. Βέβαια, πάντα παραμένουν τα θέματα τα εκκρεμή, δεν έχουμε καταλήξει σε όλα σε συμβασμούς και πρέπει να τα συζητήσουμε. Για τις σορευτικές συνέπειες θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και θα συμπληρώσω το εξής, ότι είναι καλό βεβαίως να συζητούμε για εμπορικές συναλλαγές. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ωστόσο να εξισωθούν κατά κάποιο τρόπο, να εξισορροπηθούν διαφορετικές φιλοσοφίες ακόμη παραγωγής. Αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει Πολλές φορές βάζουμε υπερβολικές απαιτήσεις ε, στη βαλίτσα και ε, απογοητευόμαστε, αισθανόμαστε δυσφορία όταν ε, δεν ακολουθούν οι άλλοι γιατί δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές παραγωγής και βλέπουμε ότι οι δικές μας προδιαγραφές μας ισοδυναμούν με μεγάλο βάρος στην αποσκευή. Γι' αυτό λοιπόν Θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιος ε, θα κατηγορηθεί ως αποδεπουμπέος τράγος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ρίχνουμε ψόγο δεξιά και αριστερά. Είναι καλό αφενός με, να δούμε ότι η κοινωνία από τη μία μας ε, ζητά να εισαγαγούμε στο των υψηλέ προδιαγραφέ, ενώ από την άλλη βγαίνουμε στις διεθνείς αγορές και καταρρύπτουμε οτιδήποτε ισχύει ως προδιαγραφές. Ευχαριστώ πολύ. L'oiseau. L'oiseau. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διαπόστοση καταρχάς, διαπίστωση καταρχής. Ε, μου φαίνεται αντιφατικό το να θέλουμε να ανοίγουμε καινούριε αγορέ ενώ ζητούμε όλο και περισσότερη προστασία. Χρόνια τώρα εμείς ζητούμε αυτή την προστασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση του κανόνε των ελεύθερων συναλλαγών ε, την απορρίπτει. Μάλιστα υπάρχουν κράτη που απειλούνται με πρόστιμα όπως συμβαίνει με τη Γαλλία ε, για παραβίαση των συνθήκων των ελεύθερων συναλλαγών. Η Εντερμαχσέ, το, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, βρέθηκε λοιπόν ε, να λογοδοτεί γιατί θέλησε να υποστηρίξει τον τομέα του χειρίου κρέατος η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να μην είναι σε θέση η ίδια να εφαρμόζει τους κανόνες της ωστόσο μέσα στην ίδια της την αγορά και εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή, τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα με τις ε, συμφωνίες για τις οποίες γίνεται τόσος λόγος τον τελευταίο καιρό. Γίνεται προσπάθεια να μειώνονται οι εισαγωγές, ε, να προστατεύονται οι εθνικές παραγωγές των άλλων κρατών. Έχουμε να κάνουμε με ένα τρόπο, κατά έναν τρόπο με ένα κοινωνικό ντάμπινγκ το οποίο θα τις εκκίνδυνο το γεωργικό τομέα. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Ντες. Πρόεδρε, να σας πω. Μόλις το πρωί έφαγα μια μπανάνα που δεν παρήχθη στην Ευρώπη. Τώρα, τώρα πίνω έναν καφεδάκο, τον οποίο επίσης δεν έχουμε παρασκευάσει, δεν έχουμε καλλιεργήσει στην ε, Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα θετικά των ε, ευρωπαϊκών ε, εμπορικών σχέσεων με άλλες χώρες και θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ συγκεκριμένα τις ε, προτάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τον πεζορισμό φερρυπίν των τιμών. Έχουμε ένα παράδειγμα με μείωση της τιμής στο κιλό της παράνας από τα 2,75 στα 2,5 δολάρια το ευρώ για τον παραγωγό στη Βραζιλία ή σε άλλες ε, χώρες Λατινικής Αμερικής που δεν επιτρέπουν ε, τον, την επιβίωση του παραγωγού. Ε, στις αμερικανικές αγορές ήταν ε, στο σούπερ μάρκετ η τιμή 7,5 δολάρια. Στην Ευρώπη ερχόταν με 8,5 δολάρια στο σούπερ μάρκετ την μπανάνα. Πρέπει λοιπόν ε, με αυτό το παράδειγμα να δείξω ότι χρειάζεται να εισαχθούν ισότιμες συνθήκες και για τον παραγωγό. Η παραγωγή του Μερκοσούρ και θα το θυμούνται ίσως οι συνάδελφοι είχαν πολύ συχνά επισημάνει το πρόβλημα και λέγαμε ότι θα πρέπει οι γεωργικές ε, εισαγωγές να επιτρέπονται με τους όρους όμως της στήρησης, της προστασίας της κοινωνικής, της οικολογικής, της περιβαλλοντικής προστασίας των ζώων ε, και με προδιαγραφές βέβαια παραγωγής αντίστοιχες με τις δικές μας. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ισότιμο εμπόριο. Για δε τα ευαίσθητα και τα προϊόντα, θα πρέπει να κοιτάξουμε τους όρους υπό τους οποίους θα έρχονται από τη Λατινική Αμερική, από τη ε, τα προϊόντα αυτά στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πιο δυσμενείς συνθήκες στους δικούς μας γεωργούς και πάνω απ' όλα δεν μπορούμε να τους ταλαιπωρούμε με υπερβολικές γραφειοκρατικές ε, επιβαρύνσεις όπως συνέβη με έναν γεωργό της δικής μου περιφέρειας ο οποίος επειδή για 14 μέρες ήταν άρρωστος και δεν μπόρεσε να κάνει τα γραφειοκρατικά ε, που προέβλεπε η νομοθεσία επιβαρύνθηκε με 6.000 ευρώ πρόστιμο ε, κάτι το οποίο φυσικά δεν απασχολεί ποτέ έναν Βραζιλιάνο καλλιεργητή. Αλλά δεν δεν είναι κανείς από τους πράσινους <coughs> για να λάβει το λόγο. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ. Εδώ και πολλή ώρα ε, μιλούμε και εδώ και πολύ καιρό μιλούμε για την κρίση στο γεωργικό κλάδο, αλλά την κρίση αυτή μπορούμε να την επιλύσουμε μόνο με το άνοιγμα νέων αγορών. Βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε υπερπαραγωγή, έχουμε πλεόνασμα παραγωγής και δεν έχουμε διέξοδο δεν έχουμε αγορέ για να διαθέσουμε τα προϊόντα Μα. Χρειαζόμαστε λοιπόν κατεπηγόντω νέε αγορέ. Και αυτή η συμφωνία τη που μερικοί την κατηγορούν και πολύ ποιότερα σχέση με το παρελθόν, μα δίνει ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανοίγει την Αμερικανική αγορά που μπορεί να απορροφήσει μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί φυσικά με τις προδιαγραφές ποιότητας και εκεί θα πρέπει να είμαστε ανυποχώρητη. Επίσης για τα δημητριακά, τα σιτηρά για το κρέας. Θα πρέπει να προσέξουμε και να δούμε πού θα βρούμε διεξόδους. Ε, ενώ έχουμε κλειστεί την ε, ρωσική αγορά, δεν μπορούμε να κλείνουμε τις πόρτες ε, και προς άλλες αγορές. Οι γεωγραφικές ενδείξεις φυσικά είναι κόκκινη γραμμή. Είναι ιερή και απαράβατη αρχή. Ο καταναλωτής δικαιούται να γνωρίζει την προέλευση των προϊόντων που αγοράζει. Χρειάζεται λοιπόν η χνηλασιμότητα. Και για όλες αυτές τις αρχές ε, θα μπορούμε, με σεβασμό όλων αυτών των αρχών, μπορούμε παρόλα αυτά να αναζητήσουμε νέες αγορές. Δεν μπορούμε να μένουμε εκλοβισμένοι στις παραδοσιακές αγορές. Δεν θα μας οδηγήσει πουθενά μια τέτοια κατάσταση και μια τέτοια απομόνωση. Χθες είχαμε διάσκεψη κορυφής στο Ανόβερο που επιβεβαίωσε την σκοπιμότητα της διατήρησης των κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θεωρώ ότι το άνοιγμα νέων αγορών είναι μεγάλη σημασία στο σημερινό πλαίσιο κρίσης του γεωργικού τομέα. Καλώς ξεκινούν διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, αλλά θα πρέπει να είναι ισορροπημένες στην ε, εξέλιξή τους για να έχουμε την κατάλληλη προστασία των πλέον ευάλωτων τομέων. Θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει να αρνηθούμε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση όπου η Ευρωπαϊκή Γεωργία θυσιάζεται και χρησιμοποιείται ως νόμισμα στην αγορά ισοτομιών και υπάρχουν δασμολογικέ παραχωρήσει που λειτουργούν ει βάρο τη γεωργία για να πετύχουμε τι εμπορικέ αυτέ συμφωνίε. Θα πρέπει αυτέ να πετυχαίνουν όρου ανταγωνισμού ισότιμου μεταξύ των εταίρων και των διαφόρων εμπειρευομένων στον γεωργικό κλάδο. Διότι το υψηλό κόστο που πρέπει να καταβάλουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί για την περιβαλλοντική προστασία και την επιστημιστική ασφάλεια αλλά και τι κοινωνικέ ε, πτυχέ είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να μπορέσουν να ωφεληθούν όσο γίνεται περισσότερο και οι Ευρωπαίοι Γεωργοί από το άνοιγμα αγορών. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Τζουφρίντα ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να είναι συνεκβανών προπόθεση για, την, ε, για τις διαπραγματεύσει μα, τι εμπορικέ συμφωνίε με τρίτε χώρε. Ιδίω για αυτέ που έχουν προβλεφθεί ήδη ε, στο πλαίσιο του TTIP. Ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τον κύριο Νταντά τις ε, καταληκτικές παρατηρήσεις, αν φυσικά το επιθυμεί. Δεν είναι υποχρεωτικό. Σημειώσαμε μαζί με τη βοηθό της κυρίας Σαράς Γκαρσία όλες τις παρατηρήσεις ε, των συναδέλφων και θα τις μεταφέρω πιστά στην εισηγητριά μας, την κυρία Εράς Γκαρσία, μαζί με το περιεχόμενο της συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να στείλουμε επιστολή στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, γιατί για το σημείο αυτό δεν βλέπω κανέναν εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι, αλλά για άλλα σημεία αρμόδια, όχι για το συγκεκριμένο σημείο. Θα διαμαρτυρηθούμε λοιπόν. Θα στείλουμε σχετική επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έστειλε για το σημείο αυτό εκπρόσωπο και να κάνω και μια παρατήρηση. Φυσικά το ελεύθερο εμπόριο ε, πρέπει να είναι επωφελές για όλους. Αλλά ε, να διαφυλαχθούν οι αρχές του θεμητού ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα αυτό στις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει στις διαπραγματεύσεις να ληφθούν υπόψη και τα ειδικά συμφέροντα των επιμέρους κλάδων και να δώσουν την ευκαιρία για αμοιβαίο ε, όφελος. Να μην είναι ετεροβαρής μόνο υποχρεώσεις. Επίσης, κάποιος θα πρέπει να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των γεωργών. Γιατί αν είναι αρνητικά τα αποτελέσματα, κάποιος θα πρέπει να τους αποζημιώσει για τις αρνητικές συνέπειες τέτοιων εμπορικών συμφωνιών. Επίσης, θα πρέπει να μεταφέρουμε την απόφαση και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφή ε, του Ανοβέρου ήταν ομόφωνη η απόφαση για παράταση των κυρώσεων ε, προ τη Ρωσία. Εντάξει, καταλαβαίνουμε την πολιτική σκοπιμότητα, αλλά μην ξεχνάμε και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων Γεωργών που θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Επίσης, ε, μανιωδώ επαναλαμβάνω και θα με περάσετε και για ιδεολειπτικό, Έφυγε η κυρία Μαγκίνε στο μεταξύ, αλλά θα πρέπει αντιπρόεδρος ε, να μεταφέρει αυτά τα θέματα και στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο, στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια ξέρουμε ότι ο κύριος Σούλτς, ο πρόεδρός μας, είναι αρκετά φιλελεύθερος και ανοιχτό σε θέματα ε, ελεύθερου εμπορίου. Θα πρέπει αυτά να τα μεταφέρουμε και σε επίπεδο Προεδρείου, σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο, στο Κοινοβούλιο. Επίσης, ε, αν φτάσουμε στο αποκορύφωμα των παραχωρήσεων, θα είναι πολύ αργά για να μεταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κραυγή απελπισίας των Ευρωπαίων Γεωργών. Ε, έχουμε μέχρι τέλη Απριλίου στις 12 το μεσημέρι την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστούμε την κυρία Μαγκίνες την, την κύριο συγγνώμη ήταν που αντικατέστησε την κυρία Ράς Γκαρσία. Γκαρσία. Ε, ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. Ζητούμε συγγνώμη από τον κύριο Γκάιερ που τον αφήσαμε να περιμένει τόση ώρα. Αλλά δεν ήταν κακό που είχατε την ευκαιρία να ακούσετε μια τόσο σημαντική συζήτηση για την απελευθέρωση του εμπορίου. Είναι σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη με ισορροπημένο τρόπο τη γεωργία για να έχουμε πραγματικά μια βιώσιμη γεωργία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε κύριε Γκάγερ. Είστε ορμόδιο ε, εισηγητή ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών για τον προπολογισμό του 2017. όπω ξέρετε από εμά εισηγητή αρμόδιο για τα θέματα αυτά είναι ο κύριος Γιάννη. Με αυτό θα συνεργαστείτε. Πάμε στα σημεία 8 και 9 τη ημερήσια διάταξη και θα δώσω τον λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιένς Γκάιερ. Ή μήπω πρώτο τον κύριο Γιάρ. Θέλετε πρώτα. Ποιο είναι, ποιο πρώτο. Συμφωνήστε, κανονίστε μεταξύ σα ποιο θα πάρει πρώτο το λόγο. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, vielen Dank für die Gelegenheit, äh, heute Morgen Ähm, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε για μια ανταλλαγή απόψεων ως προς τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2017. Ξεκινώ με μια σύντομη παρατήρηση σε σχέση με την εξέλιξη των συνομιλιών. Ε, αναμένεται η δημοσίευση του σχεδίου προπολογισμού για το 2017 από την Επιτροπή στις 25 Μαΐου, οπότε και ξεκινάει η ουσιαστική αντιπαράθεση επί της ουσίας για το, για το προσχέδιο αυτό. Προς το παρόν, τα δύο σκέλη της Μεσονομικής Αρχής, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, έχουν μόνο δύο έγγραφα στη διάθεσή τους που προσδορίζουν ε, τις κατευθυντήρες γραμμές του εκάστοτε θεσμικού οργάνου για τις ε, επερχομένες αυτές συνομιλίες. Το Κοινοβούλιο με τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες έχω καταθέσει εγώ στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και οι οποίες στη συνέχεια πέρασαν από μια πολύ επικοδομητική διαδικασία με συμπλήρωση και διεύρυνση του το Μάρτιο έχουν τη μορφή αυτή ως ε, φιλοπορίας, ως τεχνικό δελτίο θα λέγαμε για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. τις οποίες θα αναπτύξουμε και θα ε, διεξαγάγουμε εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή προς το παρόν δεν έχουμε παρά μόνο το σημείο κινήσεως για τα δύο θεσμικά όργανα που συνιστούν την ε, ε, Δημοσιονομική Αρχή, αλλά συγκεκριμένες προτάσεις δεν υπάρχουν γιατί δεν έχει κατευθεί το προσχέδιο του προπολογισμού. Πάντως, από τις διαπραγματευτικές αυτές θέσεις Συμβουλίου και Κοινοβουλίου μπορούμε να αντλήσουμε κάποιες ε, προϋποθέσεις, γενικότερες προϋποθέσεις σχεδίου για το, ε, πλαισίου για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν αυτές οι συνομιλίες. Δυστυχώς, πρώτη παρατήρηση, το Κοινοβούλιο από την σύναψη της συνθήκης της Λισαβόνας δεν είναι πια ε, στην παλαιότερη ισχυρή θέση που είχε στη διαδικασία του προϋπολογισμού, καθώς η συμφωνία η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε μέσα σε μία ανάγνωση, πράγμα το οποίο σημαίνει πως βεβαίως έχει ιδιαίτερα ισχυρή θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις προτάσεις που θα καταθέσει και τη διαμεσολάβησή έτσι μεταξύ των δύο σκελών του προϋπολογισμού και βέβαια πολύ ισχυρή θέση είναι και αυτή της Προεδρίας του Συμβουλίου. Πολύ ανάμεικτα είναι η εικόνα από την εμπειρία που είχαμε τα τελευταία χρόνια, από τη στάση της ε, των Προεδριών του Συμβουλίου και χωρίς να θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες και εις βάθος την υπόθεση αυτής, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς τη στάση και βέβαια τη δυνατότητα που έχει μια Προεδρία να εξασφαλίσει συμφωνία σε επίπεδο μελών του Συμβουλίου και μετά να πάει στο Κοινοβούλιο και να πει «Α, κοιτάξτε, μέχρι εδώ μπορούμε να φτάσουμε, ήταν τόσο λεπτή αυτή η ισορροπία που εξευρέθησε σε επίπεδο Συμβουλίου, που δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, πρέπει να την δεχθείτε όπως έχει». Βεβαίως, αυτή είναι η εμπορία που είχαμε στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα φτάσαμε μέχρι το σημείο σκεφτόμαστε ότι μας έχουν φέρει εδώ πέρα για να επικροτούμε μόνο, να δίνουμε δηλαδή ένα χειροκρότημα σε μια συμφωνία που έχει ληφθεί χωρίς δική μας συμμετοχή. Η Λουξεμβουριανή Προεδρία ε, προσδιορίσε μια διαφορετική στάση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση. Η Σλοβακική βέβαια Προεδρία έχει εν προκειμένου θέση κλειδί και χαίρο που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα το απόγευμα να δούμε τον πρέσβη τη Σλοβακία στην Επιτροπή για να ε, σε μια συνομιλία για να μπορέσω να διαγνώσω την στάση της ε, Σλοβακίας, της Σλοβακικής Προεδρίας εν προκειμένου. Από το Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, άρχισα να διαβάζω τις προτάσεις και με, διαρωτήθηκα μάλλον μήπως είχα πάρει στα χέρια μου λάθος έγγραφο. Γιατί ήταν ακριβώς ταυτόσιμο με τις κατευθύνσεις γραμμές του προπολογισμού του 2016. Το ξανακοίταξα, το ξαναματακοίταξα και είδα ότι οι τέσσερι πρώτες σελίδες ήταν ακριβώς χωρίς ούτε κόμμα να έχει αλλάξει αντιγραφή των ε, κατευθυντηρίων γραμμών του προηγούμενου έτους και μόνο μετά από αυτές τις πρώτες σελίδες γίνονται κάποιες μικροαλλαγές και φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η πλευρά του Συμβουλίου ε, μπαίνει στις διαπραγματεύσει για το 2017 με μια ε, πρακτική με μια θέση απαράλλακτη σε σχέση με αυτή του προπολογισμού του 2016. Όπου είδαμε πως η προσέγγιση της Επιτροπής εν των εξελίξεων και κυρίως των κρίσεων που ξεσπούσαν χρειάστηκε να τροποποιηθούν, που ξέσπασαν μάλλον το μεταξύ, χρειάστηκε να τροποποιηθούν ριζικά και στην εσωτερική πολιτική και στην κατηγορία 4 με την εξωτερική πολιτική χρειάστηκε να αλλάξει το περιθώριο που είχαμε στη θέση μας με τα ανώτατα όρια για τον προπολογισμό, για το μεσοπρόθεσμο μεσονομικού πλαίσιο επίσης τα μεσοπρόθεσμα τα ανώτατα όρια, χρειάστηκε να αλλάξει η κατάσταση να απορροφήσουμε το δυνατόν ε, τα κονδύλια που είχαμε στη θέση μας ακόμη και με τα περιθώρια γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση σε ενδιάμεση φάση με την κατηγορία 4 δηλαδή αξιοποιήσαμε, απορροφήσαμε όλα τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ε, απειλές και τα προβλήματα και επίσης να βοηθήσουμε τα ε, κράτη που βρίσκονται στην πολύ εγγυή γειτονία μας όπως η Συρία. Στην κατηγορία 3 λοιπόν, στην ιστορική πολιτική κοινοτοποίησαμε κάθε μέσο που είχαμε στη διάθεσή μας προκειμένου να στηρίξουμε τα κράτη που ε, αντιμετωπίζουν τις συνέπειες προσφυγικής κρίσης. Το περιθώριο δηλαδή είναι μηδενικό. Το δε συμβούλιο μπαίνει σε πραγματικά διαπραγματεύσεις λέγοντας αμέγιστο επίπεδο το ίδιο. Περιθώριο μεταξύ ε, ανώτατων επιπέδων του του μεσονομικού πλαισίου και του συνολικού προπολογισμού. Αυτά δηλαδή και το μεσοπρόθεσμων προοπτικών, συγγνώμη. Ε, άρα το, το Συμβούλιο δεν κάνει καμία νέα πρόταση, δεν προσπαθεί καμία νέα λύση να δώσει. Ε, βρίσκεται σε μια καταγραφή στιγμιότυπου μόνο, στιγμής δηλαδή, και η Επιτροπή καλείται να ε, εκτελεί τις πληρωμές της με βάση κάποια κριτήρια τα οποία θα σημαίνουν πως θα πρέπει να αναζητεί με τον πιο ευφύ τρόπο τα προγράμματα στα οποία δεν θα υπάρξει επαρκής απορρόφηση, όπου ε, ίσως θεωρεί το Συμβούλιο ότι θα είναι τόσο χρήσιμο για να απορροφηθούν τα, κριτήρια, τα, τα κονδύλια, ώστε από εκεί να μεταφέρει ποσά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τα αξιοποιήσει εκεί που χρειάζεται. Και το θέμα είναι ότι εμείς ως Κοινοβούλιο δεν έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τα σημεία, τα κέρια του προπολογισμού, στα οποία θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Τα δύο τρίτα του προπολογισμού τα είδαμε ε, με τις κατευθύνες γραμμές που εγκρίναμε το Μάρτιο στην Ολομέλεια και νομίζω ότι από τις συνέπειες των κρίσεων που είχαμε αναγνωρίσει ήδη το 2015, στα τέλη του 2015, δεν βλέπουμε να έχει εξεφανιστεί καμία, παραμένουν όλα τα προβλήματα ανοιχτά ε, και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις συνέπειες της ε, προσφυγικής κρίσης η οποία θα συνεχίσει και φέτος και του χρόνου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα τελειώσει. Η οικονομική κατάσταση παραμένει η ίδια. Είναι ακόμη πολλά τα προβλήματα, τα οικονομικά σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και θα πρέπει να μας απασχολήσει το πώς ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός με τα περιορισμένα μέσα που έχει στη διάθεσή του θα δώσει λύσεις στα προβλήματα αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ενεξελίξει μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 14-20 προσδιορίζει ανώτατα επίπεδα πολλά κράτη-μέλη και το δικό μου προσδιορίζοντα αυτό το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, εξέφρασαν την ικανοποίησή του ότι για πρώτη φορά οι δαπάνε Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να αυξάνονται, μειώνονται. Αυτό είχαν πει. Και τώρα έχουμε πολλέ, πολλαπλέ κρίσει εν εξελίξει και διαπιστώνουμε ότι αυτό το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο είναι αυτό που λέμε στα, στην πατρίδα μου, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έχουμε προβλήματα στην, στο οικονομικό επίπεδο, στην μεταναστευτική κρίση, στην προσφυγική κρίση, δε, στα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσει. Πάντα χρειάζεται ένα συμπληρωματικό προπολογισμό για το 2016, το οποίο πρέπει, στον οποίο πρέπει να δώσουμε απαντήσει με επιπλέον μέσα. Το Συμβούλιο λοιπόν τι έρχεται και λέει, έρχεται και λέει περικόπτουμε τα κονδύλια. και πρέπει να υπάρξει επαλήθευση στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό για να δούμε αν έχουν λειτουργήσει τα πράγματα όπως τα θέλαμε και αν μπορούμε να καταλήξουμε στα συμπεράσματα, τα οποία όμως θα αφορούν το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή από το 2020 και μετά. Πράγμα το οποίο δεν επιτρέπει σε ολόκληρο το μηχανισμό να λειτουργήσει, γιατί χρειάζονται τα, μέσα αυτά, τα κονδύλια αυτά που θα επιτρέψει το μηχανισμό να λειτουργήσει. Άρα χρειάζεται κάποια λύση πιο ευέλικτη Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν από, τον ένα, από τη μια κατηγορία του προπολογισμού να απορροφούμε κονδύλια από, ε, προς την άλλη. Δεν είναι δηλαδή αλληλεπικαλυπτόμενες αυτές οι κατηγορίες. Εάν τραβήξουμε χρήματα από τη μία μπορεί τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας να θεωρούν ότι άτι ωραία τα καταφέραμε γιατί δεν χρειάζεται να μπούμε ε, τα, να τραβήξουμε χρήμα από το πιθάρι του, της κατηγορίας 2, αλλά δεν μπορούμε να τραβήξουμε χρήματα ούτε και από τις άλλες κατηγορίες. Αυτά λοιπόν είναι τα δημοσιονομικά μας. Έχουμε να κάνουμε με μια αποφασισμένη αποφασιστική αντίρα, αντίδραση και αντίσταση των κρατών μελών και πρέπει να βρούμε τις λύσεις τις δημοσιονομικές. Και επαναλαμβάνω, έχουμε μια διαρκή κρίση σε διάφορους τομείς πολιτικής, ε, πρέπει να βρούμε για το ΕΦΣΙ, για το σχέδιο Juncker, αρκετά χρήματα για το ποσό εγγύσεων, για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, γιατί δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στα 8 δισεκατομμύρια, είμαστε στα 3,38 δις και πρέπει τουλάχιστον στα 4 να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο για να μπορέσουμε να καλύψουμε το ποσό που χρειάζεται για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να δούμε από πού θα βγουν τα χρήματα αυτά από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, πώ θα αξιοποιηθούν κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να ε, διαχειριστούμε αυτέ τι κρίσει και με βάση βέβαια τι επιλογέ τη πολιτικές και τη... το, ιδιαίτερο βάρο που δίνουμε εμεί ω βουλευτέ, ω κοινοβούλιο. Ο προπολογισμό επίση θα πρέπει να προσφέρει υποστήριξη στην ανάπτυξη και τι θέσει εργασία. Εν προκειμένου, οι κατευθυντηρίες γραμμές ε, του Κοινοβουλίου τείνουν να υποστηρίζουν ε, προτάσεις με οικονομικά επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομικές προοπτικές, για την ανάπτυξη, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τα κονδύλια δηλαδή που θα αξιοποιηθούν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό θα πρέπει να δίνουν λύσεις για τα προβλήματα στον στους τομείς αυτούς. Θέλουμε την καταπολέμηση της ε, φτώχειας μέσα στην στρατηγική 2000, ε, Ευρώπη 2020 είναι ρητός εντοπισμένος ο στόχος και μάλιστα της καταπολέμησης της φτώχειας των παιδιών. Έχουμε επίσης, πρέπει να το αναφέρουμε, την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την ε, μετάβαση από το ένα δημοσιονομικό πλαίσιο στο επόμενο, ένα πρόβλημα μετάβασης δηλαδή, όπου η κάλυψη είναι πολύ περιορισμένη. Είναι σαν να έχουμε μια ε, κουβέρτα κοντή, να προσπαθούμε να καλύψουμε το κεφάλι μας, αλλά τα πόδια να μένουν ξεσκέπαστα. Δηλαδή κάθε φορά έχουμε περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες για να καλύψουμε όλες μας τις ανάγκες και πρέπει πάντα με ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο να παρεμβαίνουμε για να κάνουμε τριθωτικές κινήσεις. Και πάνω απ' όλα οι πολιτικές δεσμεύσεις, υποσχέσεις που δίνει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός για το τι θα καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αγνοηθεί από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Και αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα στη διαφορά στις ε, στα κονδύλια για τις πληρωμές. Είναι σαν να λέμε ε, σε κάποιον πήγαινε ψώνισε στο σούπερ μάρκετ, σου δίνω τον κατάλογο με τα προϊόντα που θέλω να μου αγοράσεις, όλα μαζί κάνουν 100 ευρώ, λέγω εγώ σου δίνω 75 ευρώ και κατάφερε εσύ να τα αγοράσεις όλα. Αυτό κάνουν τα κράτη-μέλη με τη διαφορά ανάμεσα στις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές. Και γι' αυτό νομίζω ότι Πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση και περιμένω να ακούσω και τις, τα δικά σα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Γκάιερ για αυτές τις αγωγικές παρατηρήσεις. Υπάρχει ένα ρητό πολύ, όσο πιο πολύ πλησιάζει στο γίγαντα, τόσο πιο μικρό σου φαίνεται. Εγώ νομίζω όμω ότι συμβαίνει το αντίστροφο με τον προπολογισμό. Όσο πιο κοντά έρχεται η ώρα του προπολογισμού, τόσο μεγαλύτερα φαίνονται τα προβλήματα. Έχουμε αυτή τη δυσαρμονία στην αξιολόγηση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τη σοβαρότητα των προβλημάτων που εντοπίζουμε και βέβαια υπάρχει ανάγκη για μια σταθερότητα. Πολύ καλό ακούγεται όταν έρχεται η ώρα να εκτελεστούν οι δαπάνε, τότε τα προβλήματα ακριβώ φαίνονται πολύ μεγαλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια τεράστια οικονομική κρίση στο γεωργικό τομέα, στο γάλα, στο χείριο κρέας. Έχουμε πολύ χαμηλές τιμές ε, στα σιτηρά, πρόβλημα ως προς τα εισοδήματα των γεωργών και χρειάζεται για τη σταθεροποίηση αυτών να υλοποιηθούν οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Φυσικά δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η γεωργία, ο γεωργικό τομέα και ω ε, παράγοντα τη οικονομία και ω τομέα τη οικονομία και ω παράγοντα δημιουργία θέσεων εργασία. Ήδη βλέπουμε ότι στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό οι πληρωμές του δεύτερου πυλώνα για τη γεωργία μειώνονται σε σχέση με την υπόσχεση δηλαδή, που είχε δοθεί από το Συμβούλιο ότι θα δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία κτλ., βλέπουμε ότι υπάρχει σαφώ αντίθεση. Έρχεται και μειώνεται αυτό ο δεύτερο τομέα, τα προγράμματα, τα περιβαλλοντικά, των επενδύσεων, τη καινοτομία, εκεί όπου έπρεπε να υπάρχει το αποθεματικό για την περιφέρεια, για το γεωργό, για να υποστηριχθεί. Παρουσιάζει ξεκάθαρη μείωση, πράγμα αντιπαραγωγικό και θα το επισημάνουμε φυσικά. Και επίσης είδαμε στην προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο τον ε, αποπληθωριστικό παράγοντα είχε επεκταθεί σε όλους τους τομείς του προπολογισμού πλην της γεωργίας. Τώρα βλέπουμε και στη γεωργία ορατές πλέον αυτές τις περικοπές στον προσεχή προπολογισμό. Εμείς λοιπόν θα ετοιμάσουμε τη γνωμοδότησή μας για τον συνάδελφο από την Επιτροπή των Προπολογισμών και θα υπογραμμίσουμε εκεί τη σημασία της γεωργίας ως τομέα της οικονομίας. Δεύτερο, την αντίθεσή μας ως προς τις περικοπές ε, για, το, για την ύπεθρο γενικότερα με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Και τρίτον, θα ε, επισημάνουμε πως υπάρχει οικονομική κρίση, ιδιαίτερα στο τομέα της γεωργίας, κρίση στην οποία χρειάζεται να δοθούν λύσεις. Και για να συνοψίσω, η δική σας η ε, περίληψη των προτάσεων είναι καλή, τη βρίσκω θετική και πιστεύω ότι μπορούμε με τις προτάσεις μας να υποστηρίξουμε ένα τον άλλον. Και εγώ αισθάνομαι δυσφορία ως προς το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη ζητούν πάντα να αναλαμβάνονται δεσμεύσεις, αλλά όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής δεν δηλώνουν το παρόν. Και σε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναπτύξει μια βασική γραμμή για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Έχουμε ήδη περιγράψει το φαινόμενο που είχαμε πάντα καθυστερήσει τις πληρωμές και τρέχαμε να προλάβουμε τις ε, εκρεμίσεις. Ε, υποχρεώσεις. Έχουμε προγράμματα όμως τα οποία είναι πολυετή. Έχουμε προγράμματα τα οποία ξεκινούσαν με κάποια βραδίτα και μετά αναπτύσσουν περισσότερο τα, ε, την δυναμική τους και άρα χρειάζονται πιο εντατική εκτέλεση σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε αυτό χρειάζεται περισσότερη δέσμευση από τα κράτη-μέλη. Πολλές φορές έχουν αναλυφθεί δεσμεύσει για τα οποία τα κράτη-μέλη που καλούνται να τις εκτελέσουν ε, έχουν ξεχάσει ότι υπάρχουν και δεν προβλέπουν τις σχετικές πληρωμέ. Γι' αυτό, όπως είπατε και εσεί τρέχουμε να προλάβουμε. Πρέπει να φροντίσουμε εμεί ω Κοινοβούλιο αυτό να μην ξανασυμβεί. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε μια χαλαρή εκτέλεση, διαχείριση των δημοσιονομικών μας, του προϋπολογισμού μας, και άρα, ναι, σταθερότητα, θα ζητήσουμε με τη γνωμοδότηση γιατί στους γεωρούς ε, και στον άνθρωπο της υπαίθρου αρέσει αυτή η σταθερότητα και θα κοιτάξουμε να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα τον τομέα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χόισλινγκ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τις προτάσεις σας. Συμφωνούμε εν γέννη. Όπω είπατε δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά στην πρόταση από πλευρά του Συμβουλίου. Δεν θα υπάρχουν ε, τα κονδύλια που χρειαζόμαστε. Η κατάσταση δεν είναι καινούρια. Το είπε και εσεί, κύριε Γκάιερ. Ε, οι κρίσει δεν μειώνονται. Παλαιές δεσμεύσει δεν ε, εξοφλούνται. Και πρέπει να διερωτηθεί κανεί εν τέλει το Κοινοβούλιο πώ θα αντιμετωπίσει αυτή η κατάσταση όταν βρισκόμαστε ενώπιον μια ύποχρηματοδότηση για δεσμεύσει που αναλαμβάνουμε για πράγματα που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε, αλλά που δεν μπορούν να τηρηθούν αυτές οι υποσχέσεις. Υπάρχουν κράτη, ξεκάθαρα, υπεύθυνα για την κατάσταση αυτή και την υποχρηματοδότηση. Συγκεκριμένα το κράτος των δύο συναδέλφων που μίλησαν μόλις τώρα, η Γερμανία, η οποία αντιστάθηκε δεν είχε και με δόντια στον προπολογισμό και επέμεινε ώστε να μειωθεί ω το δυνατόν ο προπολογισμό, κύριε Γκάιερ. Πρέπει λοιπόν να καλέσουμε την ε, γερμανική κυβέρνηση, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση Γερμανίας να δει την πραγματικότητα, να συνέλθει και να αναγνωρίσει ότι δεν μπορούμε να έχουμε υποχρηματοδότηση στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Υπάρχουν σαφείς πιέσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και βέβαια την Γερμανία για νέα διαπραγμάτευση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν βλέπω άλλη λύση εγώ προσωπικώς. Έχουμε να κάνουμε με συμβαστικές λύσεις, οι οποίες όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να δώσουν κανένα αποτέλεσμα, δεν θα λειτουργήσουν. Ας ε, συμπεριφερθεί λοιπόν τελικά και μια φορά έστω το Κοινοβούλιο με σοβαρότητα και να πει δεν συμπράττουμε. Δεν πρόκειται να δοθούν λύσεις με αυτά τα ποσά και να είναι τεθειμένοι και οι συγκητέ και οι συντάκτε να πούνε δεν θα συμπράξουμε, δεν θα εγκρίνουμε εν τέλει τι προτάσεις. Βέβαια δυστυχώς κάποιο κάπου τελικά δεν είναι το πράσινο φω, ε, όπω και με το τελευταίο δημοσιονομικό πλαίσιο, που όλοι λέμε τώρα ότι δεν έπρεπε να το είχαμε δεχθεί, γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, θα είχαμε τραβήξει το φρένο νωρίτερα. Αλλά νομίζω ότι πια δεν έχουμε περιθώριο να ανεχθούμε και να δεχθούμε τέτοιες προτάσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπόθηκαν πολλά που ήθελα και εγώ να τα σχολιάσω. Απλώς ε, δύο-τρεις παρατηρήσεις. Ο προπολογισμό θα πρέπει να διατηρηθεί. Μπορεί να έχουμε κάπως λιγότερο ε, ως εκατομμύρια, αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί στη ίδιο και θα πρέπει να αυξηθούν οι επιπλέον ανάγκες της γεωργίας. Δεν είναι δυνατόν οι, θύνοντες, να, οι πολιτικοί θύνοντες να λαμβάνουν ε, αποφάσεις για κυρώσεις και να μην λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στην πράξη του ρωσικού εμπάργου λόγου χάρη. Και θα πρέπει να προστατεύσουμε και την ε, ε, παραγωγή από τρίτες χώρες. Δεν μπορεί οι γεωργοί μας να ανταγωνίζονται μη δασμολογημένα προϊόντα ενώ ήδη παράγουν εξωτερό κόστος. Κάποιοι λένε ότι ορισμένε συμφωνίε δεν θα είναι καθόλου υποφολεί. Ε, αν η Αμερικανική αγορά έχει πρόσβαση στη δική μα και πολλά περισσότερο βόλιο, εκτό και να αρχίσουμε να τρώμε περισσότερο, θα πουλάμε συνολικά λιγότερο. Κάποιο θα κερδίσει και κάποιο θα χάσει. Αλλά πάντω υπάρχει μια συνολική ψευδέστηση ότι όλοι θα κερδίσουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εκτό εάν όλοι αρχίσουμε να γινόμαστε παχύσαρκοι, εξαιρετικά παχύσαρκοι και αρχίσουμε να τρώμε παραπάνω αλλά μετά θα έχουμε άλλα διαφορετικά προβλήματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια βασική έλλειψη ισορροπία όταν ε, ζητούμε από του παραγωγού να παράγουν σε μια υψηλού κόστο παραγωγή και να ανταγωνίζονται χαμηλού κόστου εισαγωγέ. Σε άλλου τομεί αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά για κάποιο λόγο γεωργοί πρέπει να δουλεύουν ε, για ψίχουλα, ενώ άλλοι σε άλλες αλυσίδες παραγωγής ε, κερδίζουν περιουσίε Σε διαφορετικού κλάδου από τη γεωργική παραγωγή. Μερικοί κάνουν, ε, έχουν ε, ε, κέρδος εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως. Και δεν καταφέρνουν τίποτα οι γεωργοί. Είναι σαν να αυτοκτονούν με τη δραστηριότητά τους. Εδώ λοιπόν κάνουμε να κάνουμε και πρέπει να προστατεύσουμε την εμπορική μας ε, δομή. Κύριε Νόιχλ, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκάιερ. Ξεκάθαρες τοποθετήσεις σας ε, για τον προπολογισμό. Θα ήθελα ιδιαίτερα για τον κύριο Γιάρα αλλά και για σας. Στο σημείο 4 να ρωτήσω. Γίνεται λόγος για πρόσθετα κονδύλια για το τομέα του γάλακτος και του χείριου κρέατος ε, σε σχέση και με τη συνέπεια του εμπάργου. Μια απλή ερώτηση. Είναι ρεαλιστικό στους τομείς αυτούς της γεωργίας να δίνουμε επιπλέον κονδύλια. Κύριε Γιάννη, καταλαβαίνω ότι θελήσατε εσείς στην συμπερίληψη του θέματος αυτού. Το καταλαβαίνω. Αλλά ο κύριος Γκάιερ, μια και είναι εδώ, ας μας πει, θα ήταν ρεαλιστικό να δοθούν επιπλέον κονδύλια. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να εξηγήσουμε στον ε, ψηφοφόρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο συναρπαστικό στοιχείο ε, του προϋπολογισμού. Τι θα κάνουμε με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα στο γεωργικό τομέα. Και μπορούμε να συζητούμε πολλά και διάφορα θέματα, αλλά ε, μία από τις σημαντικότερες απειλές στο μέλλον, ακόμη και του χρόνου, είναι η ε, προσπάθεια επανεθνικοποίησης της γεωργικής πολιτικής ε, από πολλές χώρες εξαιτίας του αδιεξόδου ή των αδυναμιών ε, του γεωργικού προϋπολογισμού της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γίγαντας στη γεωργία και στη χρηματοδότηση, αλλά από πολιτική άποψη είναι νάνος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ω πολιτικοί ηθήνοντε θα πρέπει να είμαστε σαφεί στι απαιτήσει που έχει ο γεωργικό κλάδο από τον προπολογισμό του 2017. Οι συνέπειε ε, ε, στην ύπεθρο, η ανεργία ε, είναι και στην επιστηστική ασφάλεια είναι αναφυσβήτητες. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Ό,τι αφορά τον πολιτή σχεδιασμό, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε ο γεωργικός προπολογισμό να μην είναι άλλο στα ίδια επίπεδα, ακόμη και τα εθνικά κεφάλαια. Όπως είπα και στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Βέβαια, οι άμεσες πληρωμές θα επηρεαστούν. Φαίνεται ότι προτείνεται περικοπή κατά 1,36% και ο στόχος είναι πάνω από τα ε, επίπεδο του 2000. Θα γίνει σφοδρή συζήτηση για την πιθανή μείωση, περικοπή ή την ε, επιρροή στις άμεσες πληρωμές. Τώρα, το αποθεματικό κρίσης μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά και οι εφαρμοστικοί κανόνες θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι. Και στην εκνομοδότησή μας θα πρέπει να δούμε τι έγινε με τα αναξιοποίητα κονδύλια. Πώς αυτά τα αναξιοποίητα κονδύλια, πώς θα τα επαναφέρουμε στο γεωρικό προϋπολογισμό, να μην χαθούν. Επίσης, ε, τα συστήματα ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Παρά είναι βραχυπρόθεσμα και κοντόφθαλμα και δεν μας βοηθούν για το μέλλον, ούτε θα μας επιλύσουν μελλοντικά προβλήματα. Επίσης, υπάρχει και το θεσμικό κόστος ε, των σχεδίων. Ε, γιατί αν συνεχιστεί η ανεργία θα είναι δύσκολο το πρόβλημα ιδιαίτερα για την άσκηση ελέγχου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ευθύνε. Ε, γεωγραφικές ενδείξεις. Είπαμε ότι το θέμα αυτό θα ανατεθεί σε οργανισμό, αντί να το αναλάβει μια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσοχή λοιπόν στην αναθεώρηση και στην απόφαση. Σε ό,τι αφορά ε, ε τα θέματα τα, σχετικά με το τρόφιμα, θα πρέπει να μείνουν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Άγκρης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως ευρύτερο θέμα θα πρέπει να αναφέρουμε και το ζήτημα της ε, φορολογικής εναρμόνισης ε, και το δημοσιονομικό αντίκτυπο μιας τέτοιας διαδικασίας. Θα μπορούσε και αυτό να τεθεί ως σημείο αναφοράς. Περιμένουμε ανυπόμονα στα τέλη Μαΐου την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προβλέπουμε σε καρποφόρα συνεργασία με τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να τονίσω και εγώ πως όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που προηγήθηκαν ότι δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε τη σημασία της Γεωργίας για την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την απασχόληση, την προστασία της υπαίθρου στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης και την παγκόσμια επισκεπτική ισορροπία. Εδώ επιμένω στο γεγονό ότι ο προπολογισμό του 2017 θα πρέπει να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη τη Υπαίθρου, που καλύπτονται και τα προγράμματα leader από αυτό, ε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη τη Υπαίθρου και την ε, στήριξη τη οικονομία, που επιτρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα τη παραγωγή και των προϊόντων. Εδώ λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή την ε, μέγιστη δυνατή προσοχή το τελικό επίπεδο των ε, δεσμεύσεων που θα αναλυθούν για το Ταμείο αυτό. Και να μην ξεχνάμε και τη διακύμανση των τιμών, να σταθούμε το παράγοντα που απαιτεί δράσεις ε, αποφασιστικές και γοργές για να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές μεταλλεσσόμενες ανάγκες της γεωργίας. Εδώ χρειαζόμαστε καινοτόμα πρότυπα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διακύμανσης των τιμών στις ε, γεωργικές αγορές. Ακόμη, καλό θα ήταν να προβλέψουμε επιπλέον δημοσιονομικού πόρου για τον προπολογισμό του 2017, για το γαλακτοπαραγωγικό τομέα, για το χείριο και για τα απορροκυπηστικά, για να αμβλύνουμε τι αρνητικέ επιπτώσει τη κρίση και του ρωσικού εμπάργου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα την παρέμβαση του κύριου Γκάιερ. Ε, βέβαια, δεν είναι όλα αυτά τα θέματα από δική μας αρμοδιότητα, αλλά θέλω να πω γιατί δεν ε, ανεχόμαστε περαιτέρω περικοπές και θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε νέο χρήμα, φρέσκο χρήμα στη, στο γεωργικό προϋπολογισμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη ε, σε συγκεκριμένες χώρες μέλη έχουμε απερίμωση των αγροτικών ζωνών και μεγάλη φτώχεια. Επίσης γύρωση του πληθυσμού. Και το πλεόνασμα παραγωγής δεν μας εξασφαλίζει ε, διατήρηση αυτού του φαινομένου και μετά από 10-15 χρόνια. Δεν είναι σίγουρο ότι και στο μέλλον θα έχουμε τέτοια υπερπαραγωγή. ίσως στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα επιστηστικής ασφάλειας αν παραμείνουμε κοντόφθαρμοι στην πολιτική μας. Επίσης, οι ανεργίες στις αγροτικές ζώνες είναι διπλάσια από ό,τι στα μεγάλα αστικά κέντρα και το εισόδημα είναι σχεδόν υποδιπλάσιο σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις και αυτό με βάση σημερινού δείκτες. Οπότε προς τι να μένει κανείς σε ένα χωριό ή στην Ήπεθρο, τελειώνει το σχολείο και αφήνει το χωριό του, πηγαίνει να ζήσει σε μια πόλη ή μεταναστεύει σε άλλη χώρα. Αν δεν προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα, θα αυξηθούν οι εσωτερικές μεταναστευτικές ροές. Θα εγκαταλείπεται η και θα επιτείνεται η αστιφιλία. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, υποδομές, ε, να καλύψουμε τις κοινωνικές ανάγκες και να προσελκύσουμε επενδύσεις και στην ύπεθρο. Βέβαια, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την σοβούσα κρίση που μας ταλανίζει εδώ και 1,5 χρόνο. Παρόλο που δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να βελτιώσουμε την κατάσταση, όχι μόνο δεν τη βελτιώσαμε, αλλά επιδεινώθηκε κιόλα. Και ξέρουμε ποια είναι η αιτία της κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε και τη σωστή λύση. Να την αντιμετωπίσουμε εφαρμόζοντας ε, πιστά την νομοθεσία που έχουμε ή να προβλέψουμε συμπληρωματικέ ενισχύσει. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Δεν φταίει η γεωργία για την κρίση. Δεν φταίει η γεωργία που δημιουργήθηκε σύραξη μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία. Δεν φταίει η γεωργία, ο γεωργικό κλάδο που επέβαλε η Ρωσία το εμπάργκο. Παρ' όλα αυτά, πληρώνεται σπασμένα αυτό το εμπάργκο. Οι γεωργοί γίνονται τα θύματα. Παρόλο που δεν είναι η υπέτη της κρίσης, οι γεωργοί είναι τα θύματα της κρίσης δεν θα πρέπει να βοηθούμε μόνο ε, συγκεκριμένους τομείς με ενισχύσεις όπως το γαλακτοκομικό τομέα ή το χείριο. 3,5 δισεκατομμύρια θα βρέθηκαν για την επίλυση του προσφυγικού. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε νέο χρήμα και για τη γεωργία. Γιατί να μην εφοδιάσουμε τους καταβλισμούς προσφύγων με φρέσκα νοπά προϊόντα, τυριά, βούτυρα και άλλα νοπά γεωργικά προϊόντα. Είναι μεγάλη αγορά. Γιατί να μην βρούμε τέτοια διέξοδο για την παραγωγή μας στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Μέτρα υπάρχουν. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους γεωργούς μας, να μην τους αφήσουμε ανυπεράσπιστους. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε σημαντικό πρόβλημα και στο μέλλον. Ο κύριος Τάκουλα. Kiitoksia, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάρ πολύ καλή ισορροπημένη η γνωμοδότησή του για τις δημοσιονομικές προτάσεις για το 2017 ε, ιδιαίτερα μάλιστα υπογραμμίζει σημαντικά για τη γεωργία θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η ισορροπία στην τροφική αλυσίδα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, η παραγωγή, Και αυτά θα ήθελα να καταγραφούν με ιδιαίτερη έμφαση στην ε, γνωμοδότηση, όπως άλλωστε και το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε κάπου μια έκφραση που να μιλάει για τουλάχιστον ένα ελάχιστο. Και σε αυτό... Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις επιδοτήσεις, για το χείριο κρέας, για το γαλακτοκομικό τομέα και τους λοιπούς τομείς ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες της κρίσης. Δεν πρέπει να λησμονούμε ε, ε, την συνέπεια, μια σταθερή δηλαδή σχέση στην εισαγωγή των μέτρων αυτών. και μια συνέχεια ύστερα από την κατάρριψη των ποσοστώσεων, Φερρυπίν. που μπορούμε να θεωρήσουμε εκ των υστέρων ήταν μια καλή απόφαση. Όταν, είχαν πρωτοπροταθεί όταν είχε πρωτοπροταθεί αυτή η κατάργηση, τουλάχιστον για την πατρίδα την είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρο και συζήτηση. Τώρα βλέπουμε ότι ε, ήταν ισόφελος ε, τη γεωργία. Πρέπει πάντως να φροντίσουμε να στηρίξουμε τις πιο αδύναμες περιοχές, να αποφύγουμε την υπερβολική συγκέντρωση στα χέρια λίγων ε, της γεωργικής παραγωγής, Και γι' αυτό εγώ θα καταθέσω κάποιες μικροτροποποιήσεις, μικροτροπολογίες ε, στη γνωμοδότηση, αλλά κατά άλλα θεωρώ ότι είναι πολύ καλή εκθέση του κυρίου Γιάρ και τον ευχαριστώ. Μάλιστα, δεν έμεινε άλλο στον κατάλογο των ομιλητών. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, στον Διευθυντή, τον κύριο Χάισλερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω μόνο κάποια προκαταρκτικά σχόλια σήμερα όπως περιμένετε, γιατί στις 25 Μαΐου θα υποβληθεί επισήμως η πρόταση. Το πρώτο μήνυμα είναι το μήνυμα της σταθερότητας. Η κατάσταση προβλέψεων ε, για το 2017 ε, προτείνουν περιχαράκωση των στόχων της ΚΑΠ και των στόχων ε, της αναθεώρησης. Για το μεγαλύτερο τμήμα των άμεσων πληρωμών ήδη έχουμε δεύτερο χρόνο εφαρμογής και έχουμε μπει σε κανονική πορεία ε, σε ό,τι αφορά τα μέτρα της αγοράς, αυτό που βλέπουμε προς το παρόν για το 2017 ως πρόβλεψη είναι ίσως χαμη, κάπως χαμηλότερο από τα, δαπάνε του 2016 εξαιτία του γεγονότος ότι το πακέτο των 500 εκατομμυρίων θα έχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα στην παρούσα διαχειριστική χρήση το 2016. Λίγα θα δαπανηθούν από τον επόμενο προπολογισμό το 2017. Τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο αυτή την πληροφορία έχουμε. Για τα απορροκυπευτικά, το σημαντικό μήνυμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να παρατείνει τα μέτρα για την απόσυρση όσο κρατά το ρωσικό εμπάργο. Ένα άλλο θέμα που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην διάρθρωση του γεωργικού προϋπολογισμού για το 2017 είναι ότι εξαλείπτονται οι, οι εισφορές για το γάλα. Γιατί αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό τμήμα του προπολογισμού. Με την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων ε, εξαφανίζονται και οι σφορές ε, για το γάλα και αυτό από το 2017. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα είναι κάτω από τα ε, μεμονωμένα καταναλωτόρια του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου. Υπήρχε τέτοιο ανωτόριο για το τομέα 2. Ο γεωργικός περιπολογισμός θα μείνει κάτω από αυτό το ανωτόριο του τομέα 2 και ίσως είδατε και την πρόταση για τη δημοσιονομική πειθαρχία που θα ισχύσει μόνο για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού κρίσης της γεωργίας, μια και δεν υπάρχουν περαιτέρω ανάγκες πέραν του αποθεματικού κρίσης αυτό το στάδιο. 450,5 εκατομμύρια ήταν το προτινόμενο ποσό για το 2017. Σε ό,τι αφορά το θέμα ανάπτυξη της υπαίθρου, οι, πληρω... οι πιστές πληρωμών είναι στα όρια που προβλέπονται στα ανώτατα ε, στα πλαφό του 2017 από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε μια επικάλυψη στη με τη νέα περίοδο προγραμματισμού και σημαντικά ποσά που θα πρέπει να επιστραφούν στα κράτη-μέλη για το κλείσιμο των προγραμμάτων του προηγούμενου ε, Τη προηγούμενης περίοδου προγραμματισμού για τα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου. Βέβαια, περισσότερε λεπτομέρειε ε, ε, θα υποβληθούν στις, στα τέλη Μαΐου, 25 Μαΐου, θα υποβληθεί και επισήμως η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, περιμένουμε τους καταλόγους και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να έχουμε πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση για τα πιλωτικά προγράμματα. Αυτά ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Δευθυντά. Ο κύριος Γκάιερ τώρα και μετά ο εισηγητής μας ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Φυσικά δεν μπορώ να α, απαντήσω αναλυτικά σε κάθε τοποθέτηση. Πολλοί συνάδελφοι και σωστά σχολίασαν τη γνωμοδότηση ε, του κυρίου για αυτή είναι η δουλειά της Επιτροπής Γεωργίας. Θέλω μόνο για κάποια σχόλια να πω, εκεί όπου απευθύνονται σε μένα ερωτήσεις και που νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να δώσω κάποιες διευκρινήσεις για να συμβάλλω στη συζήτηση με αυτές. Τα εξής. Υπήρξε μια ερώτηση για το αν θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα για διεύρυνση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Φυσικά αυτό δεν το συζητούμε εμεί, ε, δεν το αποφασίζουμε εμεί στην ε, ετήσια διαδικασία του προπολογισμού, αλλά σε γύρου όπου το ζητούμενο είναι το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, άρα από 2020 και μετά. Και ως εκ τούτου τώρα λίγο πολύ ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Ήδη τα κράτη-μέλη έχουν ε, ξεκινήσει μεταξύ τους μια συζήτηση, έγιναν σεμινάρια στο Βερολίνο και το Άμστερνταμ με την Προεδρία, με την ευκαιρία της Προεδρίας, όπου πολλά ζητήματα και μάλιστα εξεπλάγει πρέπει να πω, συζητήθηκαν ε, πολύ ανοιχτά σε πολλές περιπτώσεις και ακούστηκαν κάποιες ε, ιδέες που με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι να υπήρχε η δυνατότητα να ανοίξει περισσότερο το θέμα, αλλά από την άλλη το κριτήριο κριτήριο θα είναι τι είδου προτάσει θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου. Η Επιτροπή, και δεν χρειάζεται κανεί να είναι ε, medium για να το προβλέψει, ε, θα έχει πολύ πιο επιφυλακτική ε, στάση και θα προσπαθήσει να αποφύγει το άνοιγμα συζητήσεων για τον ισχύοντα προϋπολογισμό ώστε, προϋπολογισμό, ώστε να μην θεωρηθεί ότι οι προτάσεις για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο σχετίζονται με τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό του 2017. Αυτό όμως πρέπει να το κάνουμε εμείς. Πρέπει να το ζητήσουμε εμείς και νομίζω ότι δεν θα σας ξαφνιάσω αν πω ότι πρέπει να κοιτάξουμε προσεκτικά και πάλι το θέμα της υποστήριξης της γεωργίας, το βασικό θέμα της υποστήριξης της γεωργίας και να διερωτηθούμε εάν το δημοσιονομικό σύστημα, και προσέχω πολύ τα λόγια μου, το δημοσιονομικό σύστημα της Ευρώπης είναι το σωστό και αν έχουμε επαρκείς ιδίους πόρους, που πιστεύω ότι δεν έχουμε αν έχουμε σωστό σύστημα ιδίων πόρων, ότι το 80% του όγκου του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού, ε, του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού εξαρτάται από τα εμβάσματα των κρατών μελών, Όσο δηλαδή η κατάσταση είναι τέτοια όπου τα κράτη-μέλη ανάλογα με την εσωτερική του οικονομική κατάσταση μπορούν να αποφασίσουν ε, ή με βάση και την ιδεολογική επιλογή τους αποφασίζουν ε, για το αν θα διαθέσουν τα χρήματα αυτά αλλά εμείς δεν έχουμε ιδίους πόρους τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πιο σοβαρό. Έχουμε κάνει συζητήσει σε μια εσωτερική ομάδα. Έχουμε πει ότι δεν θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση σε υπερβολικά ευρύ πεδίο ιδεών ώστε να χαθεί η ουσία. Είπαμε ότι περιμένουμε μια συγκεκριμένη πρόταση από την ομάδα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε, θα αρχίσουμε να δίνουμε τις απαντήσεις. Βέβαια, τίθεται το θέμα ε, των ε, ακόμη ανεξόφλητων ε, δεσμεύσεων, των ανεξόφλητων λογαριασμών. Βεβαίως. Έχουμε ακόμα και ζητώ συγγνώμη από τους Τσέχους συναδέλφους γιατί η έκφραση στα γερμανικά χρησιμοποιεί τον όρο τσεχικό θέατρο σκιών. Έχουμε ένα θέατρο σκιών λοιπόν στην, ε, ε, στην Γερμανία όπου ε, κάνουμε μια προσπάθεια να φτιάξουμε κάτι αλλά μετά βγαίνει ένας πρεσβευτής ο οποίο μα λέει, α, όχι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα λέει ότι έχουν παραμείνει ανεξόφλητοι λογαριασμοί και όλα αυτά δεν έχουν καμιά σημασία κτλ. Αναλύουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο, το γιογιό, το οποίο μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα μας ξαναφέρει στην ίδια κατάσταση, σοβαρές δεσμεύσεις και όχι ισοδύναμες πληρωμές. Σε μια περίοδο πληρωμών θα βρεθούμε πάλι ενώπιον των ίδιων προβλημάτων. Ο κύριος Χόισλινγκ μας μιλάει για τα συμπεράσματα στο οποία θα πρέπει να καταλήξουμε. Ναι, ακούω αυτό που λέτε, σας παρακολουθώ κατά κάποιο τρόπο. Και εγώ, σοσιαλδημοκράτης, ο κύριος Γιάρ Χριστιανοδημοκράτης, θελήσατε να επιτεθείτε κατά της συμμαχίας αυτής της πολιτικής για αυτό που κάνει και εμένα όμω στη Γερμανία με ενόχλησε το 2013 όταν μια χριστιανοδημοκρατική και φιλελεύθερη συμμαχία κυβερνητική ήρθε στο Βερολίνο για να πει «Α, ήρθε η ώρα τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει οικονομία». Οικονομία για την οποία βέβαια δεν μας έλεγε προ τα πού θα τίνει. Είναι πολύ απλό. Όσο δεν γνωρίζουμε πόσο καταρτίζεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, αυτό θα συμβαίνει. Εμένα η δουλειά μου, το μεγαλύτερο, για να μην σας πω, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου, πάση περιπτώσει, είναι να ενημερώνω τον κόσμο και τα μέσα ενημέρωσης στο τι σημαίνει ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, πού πηγαίνει ε, το χρήμα του ευρωπαίου φορολογουμένου. Και προσπαθούμε να αποφύγουμε το χειρότερο, με τα προσωρινά 12 κάθε χρόνο δηλαδή, να αποφύγουμε την πυρηνική καταστροφή, επιτρέψτε μου αυτή την ε, χονδροειδή έκφραση, ε, χωρίς όμως να λύνουμε κανένα πρόβλημα. Μπορεί ο γεωργικός τομέας να ξεφύγει από τα προβλήματα. Να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δίνω λεφτά για τη γεωργία και να πούνε και οι άλλοι τομεί, εντάξει, θα αντέξουμε να μην διατεθούν αυτά τα κονδύλια, να αντιδράσει λέει, το κοινοβούλιο έτσι, ώστε να περάσουμε σε μία διαχείριση του τύπου 12 τιμωρίων, για να μπορέσουμε μετά, ενώπιον του κινδύνου της πυρηνικής καταστραφής, να πούμε Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα, δεν λύνονται τα προβλήματα, είναι πολλά τα κοινωνικά προβλήματα στη γεωργία, δεν ε, δίνουμε απαντήσεις με τον τρόπο αυτόν. Αλλά αντέχει η γεωργία το σύστημα των δεδεκατημωρίων για ένα διάστημα. Πείτε μου το ναι και προχωράμε. Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε τις συνέπειες που θα έχει μια τέτοια επιλογή. Και ξέρω ότι η συνθήκη δεν μας έχει φέρει σε ευνοϊκή διαπραγματευτική θέση. Το επεσήμανα και εγώ ο ίδιος από την αρχή. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε με αυτό όμως και να προβάλλουμε τα επιχειρήματά μας, τα λογικά επιχειρήματα, τα επιχειρήματα λογικής που λένε ότι έτσι δεν λειτουργεί το σύστημα. Και τα κράτη που είναι καθαροί χορηγοί ας συνειδητοποιήσουν επιτέλους τι ευθύνη φέρουν. Και για την κυρία Νόχιλ που με ρώτησε εάν είναι ρεαλιστική η στήριξη που προτείνεται. Αγαπητή κυρία Νόχιλ, αγαπητή Μαρία. Η πρόγνωση, ξέρεις, η πρόβλεψη, όπως λένε, έχει το εξή μειονέκτημα ότι την ε, διαψεύδει ή την επικυρώνει το μέλλον. Τότε ναι, λοιπόν, θα μπορούσα να απαντήσω θετικά σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεχθεί να διαθέσει προς τρακονδύλια. Αν όμως αποφασίσει το Συμβούλιο να περικόψει εκεί ακριβώς όπου είναι πολύ υψηλές ε, οι πληρωμές, όπως έγινε με την περιφερειακή πολιτική πέρυσι, αυτό ε, σημείο βέβαια όπου τα κράτη-μέλη λένε ε, εάν αρχίσουν να περικόπτονται ακόμη τα ε, κονδύλια τότε εμείς δεν δεχόμαστε και δεν εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό. Και έτσι εγώ δεν είμαι σε θέση να προβλέψω αν αντίστοιχα μπορεί να δούμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην γεωργία. Και έτσι δεν μπορώ να δώσω απάντηση στη δική σου ερώτηση. Αν και δεν αποκλείεται να συμβεί αυτό. Όταν κανείς ε, μαθαίνει την τέχνη της ε, ρητορικής, ε, πρώτα απ' όλα μαθαίνω ότι πρέπει να κοιτάει να γίνεται αρεστό στο ακροατήριό του. Το έκανα αυτό μέχρι τώρα, τώρα θα πρέπει να γίνω και δυσάρεστο όμως στο ακροατήριό μου. Πρέπει να σας πω το εξή, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν έχουμε ευχερή επιχειρήματα να προβάλλουμε την υποστήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας. Γιατί έχει καταστεί η γεωργία δυσάρεστη μέχρι τώρα με πολύ υψηλέ πληρωμές, πληρωμές και ενισχύσεις που δεν έφεραν τα αναμενόμενα ε, αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορεί να έχει γίνει τυχαία. Μπορεί να ήταν πολύ περίπλοκοι οι κανονισμοί και οι διατάξεις. Άρα ως βουλευτές θα πρέπει εμείς ως Κοινοβούλιο να κοιτάξουμε να πιέσουμε προς μια απλούστευση των διατάξεων απλοποίηση των διατάξεων. Μπορεί να μην ήταν επαρκή η έλεγχη από τα κράτη-μέλη και σε επίπεδο κρατών μελών. Από την άλλη και εδώ έχουμε να κάνουμε με συνδιαχείριση και οι περιφέρειες δηλαδή έχουν την ευθύνη τους ε, για το πώς γίνεται η διάθεση των κονδυλίων αλλά και πώς ελέγχεται η διάθεση των κονδυλίων αυτών. Και μια και πολλές φορές ε, ακούω, αν και εδώ πέρα δεν είναι παρόντες, ε, στις επιτροπές που επισκέπτομαι από το ECR και το EFTD ότι α, δεν πρέπει να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν εκθέσεις ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο και την επαλήθευση της διάθεσης των κονδυλίων και ειδικά για τους Βρετανούς του UKIP θα ήθελα να πω και να μακάρι να το τα ακούσουν ότι το ελεγκτικό συνεδρίο με τις εκθέσεις του έχει πολλές φορές διαπιστώσει ότι το πρόβλημα στην εκτέλεση του προπολογισμού εντοπίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στη Βρετανία και άρα δεν είναι οι ελεγκτικές αρχές ε, της εκτέλεσης ε, του προϋπολογισμού στη Βρετανία σωστά, εξοπλισμένες δεν λειτουργούν σωστά και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πρέπει να κοιτάξουμε ωστόσο πάλι να διορθώσουμε τα προβλήματα γενικότερα στον προϋπολογισμό γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό του σφάλματος. Είναι περίπλοκοι λοιπόν οι κανόνες πρέπει να τους απλοποιήσουμε. Πρέπει ως εθνικοί βουλευτές και πολιτικοί πάνω απ' όλα ως εθνικοί πολιτικοί να κοιτάξουν τις ευθύνε που ε, αντιστοιχούν στα κράτη-μέλη, να σταματήσουμε να ενισχύουμε τις διατάξεις με ε, διορθωτικές κυρίες που απλώς έχουν επιπλέον διατάξεις και κανονισμούς, αυτό το gold plating που λέμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της υπαίθρου, είναι πάρα πολύ σημαντική για να δημιουργηθούν θέσεις εργασία Συμφωνώ απόλυτος όπω είπαν και συνάδελφοι, αλλά εάν έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί κατά τρόπο ελαττωματικό και ζητάμε να του δοθούν και άλλα χρήματα, τότε είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στην Επιτροπή Γεωργίας η κυρία Γεωργίευα μας εξηγεί πάντοτε πώς η ανθρωπιστική βοήθεια έχει αξιοποιηθεί ως πόρος αγοράς γεωργικών προϊόντων ευρωπαϊκής όμως προελεύσεως, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στους πρόσφυγες για να τους υποστηρίξουν ανθρωπιστικά κτλ. Δηλαδή μας δίνει ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και από άσχετους τομείς να ε, αποβεί ισόφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας εν γέννη. Αυτά μας λέει η κυρία Γεωργίευα, ίσως θα μπορούσαμε να δούμε χρήσιμα παραδείγματα στον τομέα, στην, ε, αντίστοιχα με αυτό. Πάντω ελπίζω ότι με την υποστήριξη όλων και τη συνεργασία όλων θα μπορούσαμε να έχουμε καλά αποτελέσματα για τον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Γκάιερ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κύριος Γιάρ με τα λάθη που ανέφερε ο κύριος Γκάιερ για το δεύτερο πυλώνα. Δεν ξέρω αν ε, ήταν υπερβολικά τα σχόλια που ακούσαμε ή στηρίζονται σε συγκεκριμένη τεκμηρίωση. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια συστηματική μείωση του αριθμού των ε, ασφαλμάτων. Ο κύριε Χόισλινγκ τελείωσε η στηριζονται σε συγκεκριμενη τεκμηριωση γιατι νομιζω οτι υπαρχει μια συστηματικη μειωση του αριθμου των ασφαλματων κυριε χοισλινγκ τελειωσε η συζητηση Εν πάση περιπτώσει, πολύ σύντομα όμως παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Αν κατάλαβα από αυτά που μας είπε ο εισηγητής, ήδη στάζει να προχωρήσει σε μια σύγκρουση, θεωρείται ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή για τη σύγκρουση. Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν προπολογισμό ο οποίος δεν καλύπτεται οικονομικά, δημοσιονομικά. Άρα δεν είναι σύνομος, γιατί αν εγώ εγκρίνω τη χρηματοδότηση κάποιου μέτρου και δεν προβλέπω τα σχετικά ε, κονδύλια, τότε εγώ είμαι παράνομος. Άρα, το να λέμε ότι άφοβα μου τώρα να τα καταφέρω ή μπορεί να προχωρήσω δεκατημόρια κτλ. Ε, δεν νομίζω ότι είναι επιχείρημα. Πρέπει να κοιτάξουμε το σοβαρότερο θέμα, όπως είδαμε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας. Και το δεύτερο, μια που έγινε συζήτηση νωρίτερα και για τις συμφωνίες Ελευθερού Εμπορίου, Ποιο βαθμό από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αντιστοιχεί σε δασμούς, σε έσοδα από δασμούς, γιατί αν συναυθεί η TTIP χάνουμε από τους δασμούς αυτούς τους εισαγωγικού. Επομένως, μήπως πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό μας και στη στάση μας για τον προϋπολογισμό. Γκάιερ, 12% των ευρωπαϊκών εσόδων προέρχονται από δασμούς. Πολύ σωστά λέτε ότι όσο περισσότερο ελεύθερο εμπόριο συνάπτεται και ελεύθερες ε, συναλλαγές ε, τόσο μειώνονται αυτά τα έσοδα. Βεβαίως το σύστημα των ελεύθερων συναλλαγών μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό νομίζω ότι ενισχύεται και το επιχείρημα ότι χρειάζεται ένα σύστημα ιδίων πόρων χρειάζονται νέοι πόροι. Όσο και αν το ελεύθερο εμπόριο αποβαίνει σ' όφελο γενικά τη οικονομία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αρκεί αυτό νομίζω. Μειώνονται τα έσοδα λόγω της κατάρρευσης των δασμών και άρα η πηγή έσοδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση συστέλλεται. Τώρα αν αυτό ω επιχείρημα θα πείσει το Συμβούλιο δεν ξέρω. Αλλά θα επισημάνω για μια φορά ότι τον προπολογισμό μπορούμε να τον απορρίψουμε μόνο εάν η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου για τους τομείς αρμοδιότητας αυτού είναι σε θέση να αναλάβει τη σχετική ευθύνη. Και πάντα βλέπουμε ότι έρχεται αυτή η θλιβερή στιγμή στη διαδικασία του προπολογισμού, στον πρώτο τριμερή διάλογο με τα κράτη-μέλη, όπου πέφτουμε πάνω σε ένα τείχο από μπετόν και από όλα οι ομάδες διερωτώνται αμάν τώρα τι θα κάνουμε και έρχεται η συζήτηση, στη συζήτηση η πρόταση για απόρριψη του σχεδίου του προπολίξιμου αλλά δεν προχωράμε παραπέρα. Γιατί άρα, γιατί εάν συμβεί αυτό δεν είμαστε θέση να στηρίξουμε τα προγράμματα στους διάφορους τομείς δραστηριότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι καταλαβαίνω την ε, δυσφορία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω. Για την ανάπτυξη της ε, Πέθρου, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να προσκαλέσετε εκπροσώπους του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί είναι πάρα πολλές οι ώρες μελετών που έχουν αναπτύξει σχέση, έχουν ε, πραγματοποιήσει σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου και νομίζω είναι σε θέση να συζητήσουμε μέσα στο θέμα αυτό. Και θα ήταν ευπρόσδεκτο νομίζω, για μένα τουλάχιστον θα ήταν πολύ καλή ιδέα να το πράξετε. Ναι. Εμείς πολύ συχνά έχουμε συναντήσει με εκπροσώπους ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Και τέτοιε πληροφορίε από τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου ακριβώ συλλαμβάνουμε. Ο κύριο γιαρ Γιάρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο-τρία πράγματα μόνο σημείωσα. Ελευθερία. Ε, ένα. Δύο. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Τρίτον. Πληρωμέ δεσμεύσει. Κύριε Γκάιερ, ξέρω ότι όλα τα ίδια λέμε, αλλά πρέπει τα κράτη-μέλη να πληρώνουν τους λογαριασμούς για τους οποίους έχουν δεσμευτεί. Ξέρω ότι τελευταία στιγμή πάντα έρχεται η στιγμή που ε, καλύπτουν τελευταία στιγμή τους λογαριασμούς στα κράτη-μέλη, αλλά ναι. εγώ ως ε, ε, βουλευτής, ως Γερμανός δεν μπορώ να δεχθώ να φτάνουμε στο ε, αμήν για να ικανοποιηθούν οι ε, υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε κάποιες λύσεις τακτικές για να αποφεύγουμε αυτά τα προβλήματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είμαστε ιδιαίτερα θερμοί υποστηρικτές της ανάπτυξης της υπαίθρου από τη γεωργία, γιατί αν δεν ασχοληθεί η γεωργία με την ανάπτυξη υπαίθρου ποιος θα ασχοληθεί. Βεβαίω υπάρχει το μείο συνοχής και πολλά καλά πράγματα έχει κάνει, αλλά θεωρεί την ύπαιθρο ως υπόλοιπο χώρο και άρα πάει χαμένο μεγάλο κομμάτι της ενασχόλησης και της υποστήριξης. Σε αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο θα την υποστηρίξει. Για τα πλεονεκτήματα νομίζω της υπαίθρου. Τα βλέπετε, είναι ξεκάθαρα, μπορεί να γίνει προσαρμογή ε, των περιφερειών. Οι, περιφερειών, οι περιφέρειες βεβαίως θα πρέπει να συμβάλλουν και να συγχρηματοδοτήσουν και να ελέγξουν τη χρηματοδότηση. Για το ποσοστό του σφάλματος. Βεβαίως γνωρίζουμε τις ε, ε, διαπιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχουν βασικά οι εξή λόγοι που είναι η διαφθορά, η απλή, ε, η απλή διαφθορά για την οποία έχουμε μηδενική ανοχή, καμία ανοχή, πρέπει με άτυγκτο τρόπο να την καταστήλουμε. Υπάρχει το, ο, σαν δεύτερος λόγος η αβεβαιότητα για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και τρίτον, τότε είναι πάρα πολύ περίπλοκο το σύστημα. Πάρα πολύ απλό. Ε, στη δική μου την περιοχή, άμα γίνει Φερρυπίνη η συγκομιδή τρει μέρε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, έχει παραβιαστεί ο κανόνα και υπάρχει πρόβλημα. Είναι ποσοστό σφάλματο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε να μην παρουσιάζεται κάθε ποσοστό σφάλματος ως διαφθορά. Αν έχουμε ένα ποσοστό σφάλματο 60% δεν είναι 60% η διαφθορά. Η διαφθορά είναι πολύ περιορισμένο. Ε, το υπόλοιπο ποσοστό είναι πράγματα που δεν θα πρέπει να έχουν γίνει έτσι γιατί κάτι διαφορετικό προβλέπουν οι κανόνε κτλ. Αλλά δεν συνιστούν διαφθορά. Άρα λοιπόν πρέπει να διορθωθούν τα σφάλματα, το ο τρόπο λειτουργία του συστήματο που οδηγεί σε σφάλματα γιατί είναι πολύ περίπλοκο και πρέπει με κάποιο τρόπο να διαφοροποιείται ο εντοπισμός ενός φάλματος από εντοπισμό ε, λάθους στους λογαριασμούς που οφείλεται σε διαφθορά. Όταν έχει γίνει παραδείγμα τη σφάλμα σε ύψος 16%, υπολογίζεται ότι έχουν διατεθεί εσφαλμένο κονδύλια 16%, αλλά κανείς δεν έχει μετρήσει πόσο είναι το πραγματικό αντίτιμο, πόσο πραγματικά έχει κοστίσει το σφάλμα αυτό και που μπορεί να μην είναι το 16% σε σχέση με το διορθωτικό ποσό. Κύριε Σκάιερ. Μα τα γνωρίζω κύριε Κιάρα, αυτό ήθελα να σας πω, πολύ σωστά τα λέτε. Θέλω μόνο να επισημάνω τόσο είναι υψηλό το ποστό του σφάλματος, η διεκδίκηση για την ε, υποστήριξη με κονδύλια της ανάπτυξης πέθρου δεν πρόκειται να γίνεται δεκτή και θα την απορρίπτουν δια με μια μονοκοντιλιά τα κράτη-μέλη ο κύριο Ιάρ. Ναι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περαιτέρω με το θέμα αυτό και τη διερεύνηση του σφάλματο, ώστε αυτή να αντικατοπτρίζει, γιατί δεν το πράττει ακόμα, την πραγματικότητα. Δεύτερον, ευχαριστώ ιδιαίτερος για τις πρώτες προτάσεις που ακούστηκαν. Υπάρχουν θετικά ε, σημεία και αντίκτυπος, πιστεύω, απήχηση θετική 4 Μαΐου νομίζω είναι η προθεσμία για κατάθεση των Α, 2, 2 Μαΐου, ακόμη πιο νωρί. 2 Μαΐου λοιπόν. Θα ενημερώσω εγκαίρως βεβαίως, αλλά κάπου μεταξύ 12 και 25 Μαΐου θα έχουμε μια συνεδρία των σκιωδών, ώστε να ε, συνεννοηθούμε να κάνουμε τις τροποποίησεις μας ε, με βάση τις τροπολογίες που θα έχουν κατευθεί και να είμαστε έτοιμοι για τον Ιούνιο και την ψηφοφορία. Ευχαριστώ βεβαίως τον κύριο Γκάιερ για την πολύ καλή δουλειά και τη συνεργασία. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ να επανέλθουμε λοιπόν ε, σε όλα αυτά που θα τα ξαναδούμε και στη συζήτησή μας με τους ελεγκτές του ελεγκτικού συνεδρίου. Σίγουρα θα φροντίσουμε να σας αποσταλούν αγκαίρες τροπολογίες στις 2 Μαΐου. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Γκάγερ και σας ευχόμαστε καλή τύχη στη σκληρή σας δουλειά. Συνειδητοποιούμε ότι θα είναι μέρος της όλης μας δουλειάς για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αλλά ελπίζουμε ότι η συζήτηση θα είναι πιο επωφελής από αυτό που αρχικά προβλέπαμε. Θα σας παρακαλέσω το απόγευμα να είμαστε στην ώρα μας όλοι. Ε, το απόγευμα έχουμε μια πλούσια συνεδρίαση μπροστά μας και έχουμε και παραπάνω χρόνο μέχρι το απόγευμα γιατί κλείνουμε λίγο νωρίτερα τώρα το πρωί. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε εδώ ακριβώς στις 3 και να θυμίσω ότι έχουμε την ε, γευσηγνωσία των παράνομων ίνων. Θα πρέπει μάλλον να τα δοκιμάσουμε για να πούμε ότι είναι χάλια. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε ως εδώ, αλλά το εστιατόριο του κτηρίου μας, του κτηρίου Γιάν, οργανώνει αυτή την γευσηγνωσία. γιατί το τελείωσε τη συνεδρίαση, τη λήξη της συνεδρίασης για αυτή τη στιγμή. Όχι, Πρόεδρε, να μην ε, φανεί ότι είναι κάτι κακό, ότι είναι κακό το κρασί. Είναι απλώς κρασί που δεν παράγεται πια στη Γαλλία. Κατά τα άλλα μια χαρά είναι το κρασί.